Colleghi, buon pomeriggio. Iniziamo i lavori di questa seduta. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζει η συνεδρίαση. Σήμερα το πρωί, στο... μετά το πέρας των εργασιών της Επιτροπής, είχαμε τη συνεδρίαση των συντονιστών, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίναμε τις εξής αποφάσεις καταλήξαμε σε συμφωνία για τη χορήγηση κάποιων εκθέσεων και κάποιων ε, γνωμοδοτήσεων που ήταν έκρεμης. Πρώτα απ' όλα, εφαρμογή της οδηγίας για την διαχείριση των αποβλήτων. Το ΕΛΚ. Γνωμοδότηση ε, της ε, Επιτροπή για τη στρατηγική πρέπει να εφαρμόσουμε για τον χάρτη δεμελιωδών δικαιωμάτων, σοσιαλιστές, ε, Φιλελεύθερη Έκθεση του 2010 για την ηθαγένεια ε, πράσινη έκθεση για την εφαρμογή του ε, κοινοτικής του 2009. Επίσης, έχουμε την ε, οδηγία για την αναπηρία, η ECR, και μία έκθεση που πήραν πάλι οι σοσιαλιστές για τα θέματα που αφορούν ε, την ε, ελευθερία του τύπου. μέχρι την επόμενη συνεδρίαση των ε, συντονιστών θα έχουμε και για, ένα, για δύο άλλα εκρεμή θέματα την απόφαση των συναδέλφων που θα υποβληθούν σε μένα. Τα θέματα των μη αναφορών επίσης είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε την επόμενη φορά όταν θα έχουμε μαζί μας το σχετικό έγγραφο. με την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων που μας απασχολούν. Τώρα, το θέμα της Παλαιστίνης. Σχέδιο ψηφίσματος φιλελευθέρων και πρασίνων. Θα προσπαθήσουν οι διάφορες ομάδες να συζητήσουν το θέμα αυτό μεταξύ τους ώστε να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία και να δούμε αν θα πρέπει να ειδήσουμε ένα έγγραφο και τι τύπου. Επίσης, πρόταση για προφορική ερώτηση στην Επιτροπή που αφορά την αναφορά 1565 κάθετο 9 εκ μέρους της ΦΕΠΕΞ. Θα ζητήσει την επόμενη φορά. Προετοιμασία των επισκέψεων που θα κάνουμε το 2011 προβλέπονταν επίσκεψη σε τέσσερις χώρες για το 2011 και είπαμε ότι η προτεραιότητά μας δεν είναι οι απλές επισκέψεις, αλλά εξεταστικές των πραγμάτων αποστολές και επιτροπές. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, επαναλαμβάνω, σε σχέση με τις απλές επισκέψεις αυροφροσύνης που μπορούμε να κάνουμε στην ε, επόμενη συνάντηση θα ξέρουμε και ποιο είναι το σχέδιο της ε, των προβλεπόμενων επισκέψεων. Αυτά ήθελα να σας πω και περνούμε τώρα στις ψηφοφορίες που αφορούν πρώτα απ' όλα τη γνωμοδότη σχετικά με, με την ε, ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους. ΙΜΚΟ. Έχουμε μόνο μία προφορική τροπολογία. Εάν δεν ζητά κανένα το λόγο, θα ήθελα να περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε σχέση με αυτή την ε, προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχουν. Άρα θα την ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνούμε τώρα στην ψήφιση της νομοδότησης υπέρ, κατά, αποχές. ατό Εγκρίνεται. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσης διάταξης. 18. 632-2008 του Ρομπέρ Μπιντρον. Είναι ο, ο αναφέρον στην αίθουσα. Όχι, θα τον ε, αντικαταστήσει ο κ. Γκριζανιεύσκη. Πρόεδρε, ε, εκ μέρου ε, τη εκστρατεία κατά τη ομοφοβία, μια πολωνική πρωτοβουλία, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που μα επιτρέπετε να παρουσιάσουμε την αναφορά μα για άλλη μια φορά σήμερα. Επειδή αφορά μεγάλο αριθμό ομοφυλοφίλων ε, και φιλογενετικών ε, κάνουμε αυτή την αναφορά που αφορά την προστασία των δικαιωμάτων ε, για την οικογένεια ε, και ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύεται από το χάρτη ανθρώπινων δικαιωμάτων αρνούνται επιστοποιητικά οικογένειακή κατάσταση, οι πολωνικέ αρχέ σε πολίτε που επιθυμούν να συνάψουν σχέση καταχωρισμένη συμβίωση με άτομο του ιδίου φύλου σε άλλο κράτο μέλο η Πολωνία είναι μία από τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν τις σχέσεις ε, με άτομα του ίδιου φύλου και δεν δίνουν δικαίωμα συμβίωσης με άτομα του ίδιου φύλου. Από τότε που μπήκε η Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί ομοφιλόφιλοι και λεσβείες βγήκαν από την Πολωνία και μπήκαν φυσικά σε σχέσεις ε, με άτομα από άλλες χώρες οι, όλες οι εθνικές αρχές ζητούν ως προϋπόθεση ε, για, τη, την ε, σύναψη συμφώνου συμβίωσης ε, να υπάρξει μια βεβαίωση ότι δεν έχουν άλλη σχέση στο παρελθόν ζητούν εν πάση περιπτώσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που πρέπει να χορηγείται από τη χώρα προέλευσης. Το πολωνικό σύστημα δεν ε, αναγνωρίζει το γάμο με άτομα του ιδίου φύλου ή την ε, συμβίωση με άτομα του ιδίου φύλου και γι' αυτό η Πολωνία δεν ε, χορηγεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ε, πιστεύουμε ότι η επιστολή που έχει ληφθεί από τις πολωνικές αρχές και που έχει προστεθεί στο φάκελο αυτού του, αυτής της αναφοράς ε, αποδεικνύει ότι πρόκειται για παραβίαση των δικαιωμάτων που αφορά την ε, γενετήσια, το γενετήσιο προσανατολισμό. Μέχρι τώρα αρνήθηκαν οι πολωνικέ αρχέ να εκδώσουν πιστοποιητικά οικογενειακή κατάσταση για άτομα που θέλουν να συμβιώσουν με άτομα του ιδίου φίλου στο εξωτερικό και στην ε, έκθεσή μας για τις οικογένειες ε, με άτομα του ιδίου φίλου στην Πολωνία το αναφέρουμε αυτό. Σε πολλές πόλεις οι πολωνικές αρχές ε, ομολογούν ότι αρνούνται τη χορήγηση τέτοιων πιστοποιητικών και έχω ένα άρθρο από το στο οποίο μία υπάλληλος τοπική σε μια κοινότητα δηλώνει ότι η ίδια έχει αρνηθεί πολλές φορές τη χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Στη Βαρσοβία πρόσφατα στις 9 Νοεμβρίου του 2010 αρνήθηκαν τη χορήγηση τέτοιου πιστοποιητικού και έχουμε συμπεριλάβει αυτή την απόρριψη του αιτήματο. Αν η Επιτροπή Αναφορών ε, εγκρίνει την ε, δική μας θέση θα μας ενισχύσει το επιχείρημά μας για το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχει σταλεί απάντηση και στην ε, Επιτροπή ε, και ε, στα Ηνωμένα Έθνη πέρυσι τον Οκτώβριο. Εμείς πιστεύουμε ότι η άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων είναι αντίθετη προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμποδίζει την ελευθερία κυκλοφορίας ε, των ατόμων και παραβιάζει ε, τα ε, δικαιώματα των πολιτών. Το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές έχει αναγνωρίσει ανοιχτά ότι πρέπει να αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα παράλληλα με τα δικαιώματα σεβασμού της οικογενειακής και ατομικής ζωής. Πρώτη παραβίαση των δικαιωμάτων Δικαιωμάτων λοιπόν των Ατόμων και το Δικαστήριο των ε, Ευρωπαϊκών Κυριοτήτων καθώς και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το θεωρούν περιορισμό της ελευθερίας κυκλοφορίας. από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ε, των ατόμων να συμβιώνουν με άτομα του ιδίου φύλου ε, και αυτό δεν μπορεί να συμβαδίζει με την άρνηση των πολωνικών αρχών. Παρότι δεν φαίνεται ε, καταρχήν να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κοινωτικών αρχών, θα πρέπει οι πολωνικές αρχές να τηρούν αυτά τα οποία επιβάλλουν οι κοινωτικές συνθήκες. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αγκιώνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ζητήσαμε από τις ευρωπαϊκές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για να εμποδίζουν την επανάληψη τέτοιων περιστατικών. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Διότι σεβαστήκατε το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σα για να μιλήσετε. Δίνω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν τώρα το λόγο, στον κύριο Κούπερ. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις πληροφορίες. Θα θέλω να σας πω ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τέτοιους περιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ξέρετε, όπως φαίνεται και από τις προηγούμενες ε, ανακοινώσεις μας ε, στην Επιτροπή Αναφορών εξετάζουμε πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των πολωνικών αρχών, τις οποίες είχαμε τη αιτήσεις στις 15 Σεπτεμβρίου του 2010 και μπορούμε να πούμε ότι όντως κατανοούμε ότι ίσως τα πολιτικά μέτρα μπορούν να έχουν σε επιπτώσεις προς τους Πολωνούς ως κοινοτικού πολίτες όταν θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Τόσο αφορά τη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία που είναι πρωταρχική σημασία για να καθορίσουμε αν ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων εφαρμίζεται εδώ και εφαρμόζονται και οι αρχές, όπως επαναλαμβάνω, όπως το δικαίωμα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και η μη διακρίσεις βάσει των σεξουαλικών προτιμήσεων και τελικά το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτικών, εκ πρώτης όψεως δεν βλέπουμε να υπάρχει άμεση παραβίαση της οδηγίας 48 του 2004, διότι όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αξιότιμα μέλη, με την οδηγία αυτή ορίζονται τα δικαιώματα για να εγκατασταθεί κάποιος και να μείνει σε μια χώρα. Δεν φαίνεται λοιπόν ότι τέτοιου είδους δικαιώματα παραβιάζονται και το αναφέρω αυτό και για τον αναφέροντα. Τώρα, η πρόθεσή μας είναι να έρθουμε σε επαφή με τις πολωνικές αρχές και να ζητήσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις για τις επιπτώσεις, τις πρακτικές αυτού του μέτρου του πολωνικού πολίθη που επαναλαμβάνω ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις αρνητικές όταν θέλει κανείς να ε, ασκήσει το δικαίωμα διακίνησής του ελεύθερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα ήθελα να αναφέρω την πράσινη βίβλο. Διότι όπως ξέρετε στις 14 Δεκεμβρίου άρχισε τη διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναγνώριση αυτού του γεγονότος. Το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα με βέας αναγνώριση ε, του γάμου στην Πολωνία δεδομένου ότι δεν προβλέπει τέτοιου είδους γάμο η Πολωνία μεταξύ ομοφύλων αλλά κυρίως έχει σχέση με το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίες των πολιτών. Βεβαίως, όταν κάνουμε αυτή την ανάλυση θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι για την ε, κοινωνική δυσύνη και το οικογενειακό δίκαιο δεν υπάρχει κοινοτικό ε, νομοθεσία για τα θέματα αυτά των συμβάσεων συμβίωσης. Θα πρέπει λοιπόν από την οπτική γωνία της ελεύθερης εκείνης να το εξετάσουμε και να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους Πολωνούς πολίτες η εφαρμογή αυτής, αυτού του κανόνα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκέριγκαν Ότεμπελτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πολωνική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τις πράξεις της διοίκησης και για τα πιστοποιητικά. που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση και το πιστοποιητικό αυτό δεν εξεδόθη γιατί δεν είναι σύμφωνο με το πολωνικό δίκαιο. Το πολωνικό δίκαιο ισχύει στο έδαφος της Πολωνίας βάσει της αρχής της εδαφικότητας και αφορά τους Πολωνούς πολίτες που μπορεί να θέλουν να δημιουργήσουν μια οικογένεια και να ζήσουν στο εξωτερικό και ο περιορισμός αυτός δεν θα πρέπει να ισχύει για τους πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, ακόμη και αν ισχύει για τους πολλούς πολίτες στην Πολωνία. Δηλαδή, ο περιορισμός αυτός θα πρέπει να περιοριστεί στην επικράτεια της Πολωνίας. Επίσης, η δυνατότητα σύναψης οικογενειακής σχέσης θα πρέπει να προσδιορίζει την κατανόμο δυνατότητα του ατόμου να το κάνει αυτό και όχι να ορίζει ε, το σε ποια χώρα μπορεί να μπει σε μια σχέση συμβίωσης ένας πολίτης. Τα άτομα που ζητούν τα πιστοποιητικά αυτά δεν παραβιάζουν το πολωνικό δίκαιο, απλώς κάνουν αίτηση χορήγησης ενός πιστοποιητικού που αφορά την κατάστασή του, την οικογενειακή του κατάσταση και τη δυνατότητά του να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης ή γάμου. Νομίζω ότι αυτή, η αρχή, ότι αυτή η πράξη παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας. Πριν από λίγα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να βρει μια νομική βάση υπέρ του αναφέροντος. Σήμερα όμως η κατάσταση φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετική και χαίρομαι που υπάρχει η πράσινη βίβλος που ανέφερε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Επίσης, η Επίτροπος Reading είναι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά, όπως είναι υπεύθυνη για τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων γιατί τα θέματα οικογενικής κατάστασης και γάμου εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Νομίζω και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό και γι' αυτό πιστεύω ότι η αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει οπωσδήποτε ανοιχτή, διότι εναρμονίζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα του οικογενειακού δικαίου Παραδείγματο χάρη να αναφέρω το διαζύγιο και τη διεθνή προσέγγιση που ακολουθείται σιγά σιγά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο οικογενειακό δίκαιο και στην εναρμόνισή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει νόημα στο να αναφερθούμε στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την Πολωνία, γιατί όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ε, επιλέξει η Πολωνία το opt-out, όμως σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ισχύει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και γι' αυτό προτείνω η αναφορά να μείνει ανοιχτή γιατί κινούμε προ μια εναρμόνιση σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να συγχαρώ τους αναφέροντες καταρχήν που υπέβαλαν αυτή την αναφορά και χαίρομαι για τις νομικές αναφορές που είναι ευρύτατες και περιλαμβάνονται μέσα. Να πω στην Κομισιόν πρώτα ότι η οδηγία για την επανένωση οικογενειών δεν εφαρμόζεται στις, αν και στην οδηγία αναγνωρίζονται ε, ως ε, συμβεί όταν ε, μετέχουν σε τέτοια σχέση. Εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα να συστήσουν οικογένεια δύο άνθρωποι του ιδίου φίλου. Οπότε αυτά που είπατε δεν αναφέρονται, δεν έχουν άμεση αναφορά. Τώρα για το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων θα έλεγα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ζητήσει να εξαιρεθεί αλλά η Πολωνία δεν έχει εξαιρεθεί σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα που επιβάλλονται από τα εθνικά δικαστήρια. Το θέμα είναι, αφορά την απονομή δικαιοσύνης. Πρώτα απ' όλα τα εθνικά δικαιοσύνη, τα δικαστήρια πρέπει να αποφαίνονται και μετά γίνεται προσφυγή στο ΔΕΚ. Πρόκειται για διάκριση. Αν διαβάσετε την επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών και από τη διοίκηση, υπάρχει δυνατότητα, εάν γίνει θρησκευτικός ή μη θρησκευτικός ή σύμφωνο συμβίωσης, να πάρετε ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Λέει όμως, και θα σας το διαβάσω αυτό το κομμάτι, τα πιστοποιητικά που παρέχονται μαρτυρούν την απουσία συνθήκων που θα συνηγορούσαν κατά τη σύναψη του θρησκευτικού γάμου και τη δυνατότητα σύναψης γάμου ε, από τους Πολωνούς ε, στο εξωτερικό συμφώνος προς το πολωνικό δίκαιο και αυτό είναι το ανησυχητικό. Οπότε η Πολωνία επιβάλλει το δίκαιό της σε άλλο κράτος μέλος και αυτό αντιβαίνει στις διατάξεις της συνθήκης. Όπως προείπαμε, ε, στερείται κάποιος το δικαίωμα να διαμένει, να σπουδάζει, να εργάζεται σε άλλο κράτος μέλος και να αξιοποιεί τα δικαιώματα που παρέχει το κράτος μέλος στο άλλο μαζί με τις ε, υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά. Έτσι λοιπόν, ένα κράτο, ένας υπήκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν έχει το δικαίωμα να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος ε, με βάση το δίκαιο που ισχύει εκεί. Έτσι λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις βλέπω ότι το πολωνικό δίκαιο λαμβάνοντα υπόψη ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να ορίζουν ποιο θα παντρεύεται και ποιο δεν θα παντρεύεται, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία. Όταν όμω πρόκειται για την ελεύθερη κυκλοφορία και την απόλαυση του δικαιώματο σε άλλο κράτο μέλο, εκεί το κράτο μέλο δεν μπορεί να επιβάλλει περιορισμού που παρεμποδίζουν την άσκηση αυτού του δικαιώματο. Τέλο, να πω ότι εύχομαι ότι καλύτερο στου αναφέροντες θα ήθελα οι πολιτικοί στην Πολωνία να έχουν επιτυχία στις μεταρρυθμίσεις που προωθούν και όπως είπε και η Λίντια, ενθαρρύνομαι από την προσέγγιση και τις δηλώσεις της Αντιπρόεδρου και Επιτρόπου Ρέντινγκ στο Κοινοβούλιο όταν συζητήσαμε για την ελεύθερη κυκλοφορία ε, μελών ζευγαριού του ίδιου φίλου. Καλό θα ήταν η πολωνική κυβέρνηση η ίδια να κάνει μια τροπολογία απλή που θα δηλώνει αν υπάρχει ε, κόλλημα από το να συναυθεί γάμος σε ένα άλλο κράτος μέλος συμφώνως προς την νομοθεσία αυτού του άλλου κράτους μέλους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Βάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά την προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου ήμουνα εισηγήτρια σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία εξ ονόματος Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Και κάτι που είχαμε εντοπίσει τότε παραμένει το ίδιο μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μιλώ για τα διοικητικά κολλήματα που δημιουργούν διάφορα κράτη-μέλη απέναντι σε ανθρώπους που προσπαθούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Πέρα από τον πυρήνα του θέματος, που δεν είναι προσυζήτηση σήμερα, είμαστε μάρτυρες σαφών ε, διοικητικών κολλημάτων σε περίπτωση ε, της Ένωσης που προσπαθούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Όπως θα μας πει και η Επίτροπος Ρέντινγκ που θα έρθει να μας ε, μιλήσει για την ηθαγένεια, Υπάρχουν πολλά διοικητικά εμπόδια που θα απασχολήσουν την, Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή αναφέρομαι εδώ σε ε, δικαστικά θέματα, τροποποιήσεις, εστίαση σε θέματα που πρέπει να αναδειχθεί η σημασία τους, ούτως ώστε να προβούν σε αλλαγές και βελτιώσεις νομοθετικές στα κράτη-μέλη. Εγώ ζήτησα το λόγο για να πω ότι θέλω και εγώ να ζητήσω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, ενώ το θέμα των διοικητικών κολλημάτων συζητείται ε, τουλάχιστον τα διοικητικά κολλήματα που αφορούν την ελευθερία των πολιτών. Ζητώ λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ο κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε κατά την άποψή μου επιχειρήματα πολύ λογικά, σημαντικά από νομικής και πλευράς και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε και η Λίδια και ο Μάικελ Κάσμαν και όπως και συμφωνώ με αυτό που είπε και η κυρία Βαλεάν. Βεβαίω. Πιστεύω όμως ότι εδώ υπάρχουν τρία προβλήματα. Τι αποδεικνύει αυτό. Ότι έχουμε μεγάλη αντίδραση στην νομοθεσία την πολωνική και αυτό δεν είναι εξαίρεση. Πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται με μεγαλύτερη μικρότερη ταχύτητα ανάλογα με το κράτος. Θα ήθελα να πω στους ε, αναφέροντες ότι είμαι αλληλέγγυος, τους υποστηρίζω και να τους πω ότι είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στην Πολωνία κάποια μέρα θα σταματήσει αυτή η κατάσταση, θα επιβληθεί η πρόοδος και οι δυνάμεις που σήμερα εμποδίζει τους πολίτες να ζήσουν ελεύθερα και όπως θέλουν, θα σταματήσουν. Κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στην κοινωνική πρόοδο. Θα ήθελα λοιπόν να πω στους αναφέροντες ότι πρέπει να υπολογίζουν στη δική μας υποστήριξη για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Εδώ είμαστε και είμαστε πάντα υπέρ όλων αυτών οι οποίοι αγωνιούν και παλεύουν για την χειραφέτησή τους και για να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ευρωπαίους συμπολίτες τους. Τρία είναι τα προβλήματα, όπως είπα. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα με εκπλήσει τότε, και θα ήθελα κάποιος να μου το διευκρινίσει, Εάν στην Πολωνία κάποιος ζητήσει ένα πιστοποιητικό κοινωνικής κατάστασης, τον ερωτούν γιατί το θέλει. Διότι στα κράτη που γνωρίζω, όταν ζητάει κανείς ε, πιστοποιητικό κοινωνική κατάσταση, το μόνο που κοιτάνε είναι να πρέπει να δουν αν είστε ανήπανδρος, παντρεμένος ή διαζευμένος. Τώρα, αν το θες για την ασφάλεια, για να ξαναπαντρευτείς, τι τους νοιάζει. Βάζουν τη σφραγίδα στο οποίο πρέπει να λέει αυτός είναι, αυτός είναι χείρος, αυτός είναι ανήπαντρος, αυτός είναι παντρεμένος και τίποτα άλλο. Τελεία και παύλο. Αυτή είναι η πρώτη μου λοιπόν έκπληξη. Διότι νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας, ένας αστυνομικού κράτους, όπου κάποιος πολίτης ζητάει ένα πιστοποιητικό κοινωνική κατάσταση και του το αρνούνται ανάλογα με το λόγο για το οποίο το ζητά. Όταν ζητάει κανείς ένα πιστοποιητικό ε, ότι έχω εμβολιαστεί, γιατί με, θα με ρωτήσει κανείς γιατί το θέλω. Η δημόσια διοίκηση αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πει ποια είναι η οικογενική κατάσταση. Τώρα, υπάρχει το δεύτερο πρόβλημα η αναγνώριση της στην Πολωνία των γάμων ή των ενώσεων που μπορούν να έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Και θα πρέπει να γίνει και αυτό το βήμα προς τα μπρος στη χώρα αυτή. Όταν δύο πολίτες, δύο άντρες, δύο γυναίκες, ένας μια γυναίκα, συνάψουν γάμο σε μια άλλη χώρα, θα πρέπει να καταγράφεται στην Πολωνία χωρίς τίποτα άλλο. Απλώς. Τώρα, όπως, αν γίνει, αν κάποιος ε, παντρεμένος Πολωνός στο εξωτερικό ή με Πολωνή, με Πολωνό αντίστοιχα ή με ξένο ε, πεθάνει, θα πρέπει να αναγνωρίσει τη νέα οικογενειακή κατάσταση του απομείνοντος η Πολωνία. Φυσικό είναι. Τώρα, οποιοδήποτε Πολωνός ή άλλος πολίτης μπορεί να έχει παντρευτεί όπου θέλει με πολωνη με πολωνο αντιστοιχα η με ξενο πεθανει θα πρεπει να αναγνωρισει τη νεα οικογενειακη κατασταση του απομεινοντος πολωνια φυσικο ειναι τωρα οποιοδηποτε πολωνος η αλλος πολιτης μπορει να εχει παντρευτει οπου θελει με οποιον θελει σε οποιαδήποτε λιχό της κοινότητας. Τρίτο, οποιοδήποτε πολίτης, άντρα ή γυναίκα, μπορεί να παντρευτεί στην Πολωνία με όποιον του αρέσει, του ιδίου φίλου ή διαφορετικού φίλου. Τρει λοιπόν είναι οι φάσει. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να μου δίνετε ένα πιστοποιητικό χωρίς να με ρωτάσετε γιατί το το θέλω. Δεύτερον, πρέπει να αναγνωρίσετε ένα γάμο που έκανα σε άλλη χώρα. Τρίτο, επιτρέψτε μου να παντρευτώ βάσει του δικαιώματος που έχω να κάνω την δική μου ε, επιλογή όσον αφορά το φίλο του ατόμου με το οποίο θέλω να παντρευτώ. Είμαστε σε μία στιγμή την οποία οι... αυτοί που θέλουν να παντρευτούν και αυτό είναι παράδειγμα της κοινωνίας μας, όλες τις κοινωνίες είναι οι ιερείς και ομοφιλόφιλοι για να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι άλλοι πολίτες. Γι' αυτό, τελειώνοντας όπως άρχισα, θα ήθελα να πω το εξής. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τους αναφέροντες. Έχω την εμπιστοσύνη ότι θα ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες και βεβαίως δεν θα πρέπει όταν Γνωρίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Σε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης παρεμφερείς με αυτή που δεν την ξέραμε ότι συμβαίνουν, να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να αναλάβουμε δεσμεύσεις, να συνεχίζουμε τις πιέσεις μας, ώστε να εξομαλυνθούν οι καταστάσεις αυτές και να μπορούν όλοι οι πολίτες να ασκούν ελεύθερα τα θελεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σενσέν. Ε, Należy zwrócić uwagę, że odmowa wydania e, Ευχαριστώ. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η άρνηση χορήγηση πιστοποιητικού υγειονομική κατάσταση σε Πολωνού πολίτε που είναι ομοφυλόφιλοι, περιορίζει τα δικαιώματα και αυτού του ατόμου αλλά και των πολιτών από άλλες χώρες διότι το καθιστά δύνατο για αυτούς να μπουν σε σχέση συμβίωσης με Πολωνούς πολίτες αν η άρνηση είναι προς πολίτες άλλης χώρας δηλαδή που θέλουν να μπουν σε συμβίωση με Πολωνούς πολίτες άρα είναι μια διάταξη που αφορά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νομικέ διατάξει δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένε στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί τέτοια πιστοποιητικά δίδονται σε άτομα που είναι ετεροφιλόφιλοι, χωρίς να υπάρχει δυσκολία. Άρα, εδώ υπάρχει διακριτική μεταχείριση κατά των ομοφιλοφίλων. Και είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τους Πολωνούς πολίτες, αλλά και τους πολίτες όλων των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Πολωνία υπάρχει ομοφοβία. Και εμείς θα πρέπει να αντισταθούμε όπως αντιστάμεθα ε, κατά όλων των μορφών φοβίας. Ο κύριος Μποτσινάρ. Αγαπητοί. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσει. Εδώ πρόκειται για βασικές θεμελιώδεις παραβιάσεις είτε στο κράτο μέλο είτε στην Ένωση, είτε εκτό αυτή πρέπει να υπάρχει σεβασμό για θεμελιώδη δικαιώματα. Εδώ υφίσταται διακρίσεις μια ομάδα ατόμων αποκλειστικά πάνω στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού. Σε μια σύγχρονη εποχή, κανένα κράτος δεν μπορεί να δέχεται ένα κράτος μέλος αν ένας κανόνας δικαίου εφαρμόζεται ανάλογα με τη θρησκεία στην οποία ανήκει κανείς, ή το φύλλο ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Υπάρχει εδώ σαφή αντίφαση σε ένα θεμελιώδε δικαιώματα. Επίσης η εξοεδαφικότητα, η ετεροδικία, αυτό είναι το δεύτερο σημείο παραβιάσεων. Το πολωνικό κράτος δρά εκτός επικράτειά του. Έτσι, η ετεροδικία ή η εξοεδαφικότητα θεωρείται ως ανωτέρα βία σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Ούτε σε διμερείς συμφωνίες μπορεί να ισχύουν αυτά. Ότι δηλαδή θα εφαρμόζεται η ετεροδικία. Τέλος. Εδώ μιλάμε για τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, είτε στην Πολωνία είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Πολωνία θα πρέπει να σκεφτεί το ενδεχόμενο να προσυπογράψει τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να παραμείνει λοιπόν ανοιχτή η αναφορά και ελπίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει με κάποιο τρόπο να περάσει ένα στεναρό μήνυμα προς την Βαρσοβία ώστε να τροποποιηθεί η νομοθεσία και να προσαρμοστεί το περιεχόμενο του νόμου στο έτος και στην εποχή που ζούμε το 2011 όπου δεν έχει θέση η διάκριση στην Ευρώπη, τουλάχιστον θεωρητικά, τουλάχιστον στο γράμμα του νόμου. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ζήτησε το λόγο. Θέλω μόνο να σχολιάσω κάποια σχόλια που έγιναν Καταρχήν για την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία. Ακόμα και αν βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση, όπως είπα πριν, τα στοιχεία δεν καταδεικνύουν άμεση παραβίαση της οδηγίας, όλοι σας αναφέρατε την αρχή της ελεύθερης διακίνησης, κυκλοφορίας και βέβαια η οδηγία εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο σε ζευγάρια διαφορετικού φύλου όπως και σε ζευγάρια του ίδιου φύλου. Δεν προβλέπει διακρίσεις και στηρίζεται στον χάρτη ιδεολογική σκέψη της οδηγίας υπαριθμών 41 αναφέρεται ότι η εφαρμογή της οδηγίας στηρίζεται στο άρθρο 21 που απαγορεύει κάθε διάκριση με, με βάση τον γενετήσιο ε, προσανατολισμό. Επίσης, η εφαρμογή της οδηγίας δεν ε, ε, απαιτεί αμοιβαία αναγνώριση από τα κράτη-μέλη, αλλά έχουμε τις τρεις φάσεις, όπως είπατε, που απαριθμούνται, όπου απαριθμούνται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Αυτό αφορά και την Πολωνία. Πρώτον, θα είναι καλό να δούμε αν το πολωνικό μέτρο μπορεί να καταργηθεί ώστε να υπάρχει καλύτερη ε, διασφάλιση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας. Ίσως ε, πολλοί Πολωνοί έχουν ζήσει πολλά χρόνια σε ένα άλλο κράτος μέλος και θέλουν να παντρευτούν ή να συνάψουν σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης με κάποιον, ανεξαρτήτως φίλου. Το, αυτό να αναγνωρίζεται. Επίσης, σε δεύτερο στάδιο, το δεύτερο βήμα, να αναγνωρίζονται οι νομικές συνέπειες αυτής της σχέσης οι φορολογικές συνέπειες αυτής της σχέσης των ζευγαριών που έχουν συνάψει γάμο ή καταχωρισμένη συμπίωση σε άλλο κράτος μέλος και που θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα αυτά στην Πολωνία όταν ασκήσουν το δικαίωμά τους να εγκατασταθούν στην Πολωνία βάσει της ελεύθερης κυκλοφορίας. Τρίτον, αλλά βέβαια εδώ δεν υπάρχει ενωσιακή αρμοδιότητα για να επιβάλλει αυτό το βήμα, η Πολωνία να επιτρέπει στους πολίτες της να συνάπτουν ε, γάμους ή καταχωρισμένη, σχέση καταχωρισμένη συμβίωσης με άτομα του ίδιου φύλου. Βέβαια, τώρα στο δεύτερο και τρίτο στάδιο δεν έχουμε άμεση αρμοδιότητα. Η Πολωνία θα πρέπει να διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή υπηκών της Ένωσης στο έδαφος της, στα πλαίσια της ελεύθερης κυκλοφορίας και να ε, το περιορίζει μόνο με βάση κάποιους φορολογικούς λόγους. Πάντα ε, σύμφωνα με τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αποτελεί ε, ενωσιακή νομοθεσία. Τώρα, οι άλλοι τομεί του δικαίου και οι άλλες προτάσεις που ετοιμάζονται ή την χάνουν επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκατε στο εφαρμοστέο δίκαιο για το δίκαιο διαδοχής, συζυγικά δικαιώματα, δικαιώματα επί της ιδιοκτησίας και περιουσίας όταν υπάρχει καταχωρισμένη σύμβαση. Όλα αυτά στηρίζονται στο άρθρο 21 της, ε, του χάρτη και σε αυτά τα πλαίσια λαμβάνουμε πολύ σοβαρά το θέμα αυτό. Πάντα δηλαδή λαμβάνεται αυτό υπόψη όταν προτείνουμε νέα νομοθεσία για να προωθήσουμε με τρόπο θετικό τις διατάξεις του χάρτη. Ένα τελευταίο σχόλιο Υπάρχουν πληροφορίες ότι έγινε μια ανάλυση νομική επί αυτής της αναφοράς ήδη, την οποία ανάλυση όμως δεν έχω. Δεν είναι η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή που εννοώ, αλλά είναι η ανάλυση της Επιτροπής ή κάποια ανάλυση που ζητήθηκε από τον αναφέροντα και η οποία αναφέρθηκε ήδη. Αυτή είναι μια πληροφορία που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου. Θα ήθελα παρακαλώ να ξέρω, εφόσον είναι ε, δημόσια η ανάλυση αυτή, να την λάβω και να τη λάβω υπόψη μου κατά την ανάλυση αυτής της ε, υπόθεσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κάσμαν ένα λεπτό. Συντομότατος θα είμαι, κυρία Πρόεδρε, να πω ότι απογοητεύτηκα από την απάντηση της Κομισιόν γιατί στα πλαίσια του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ε, ε, ε, βεβαίως γίνονται σεβαστά και άλλα δικαιώματα, αλλά όταν δεν λαμβάνονται υπόψη θέματα ε, κράτους δικαίου με βάση το άρθρο 6, το θέμα είναι σοβαρό. Δηλαδή το, υπάρχει το, ε, η άρνηση του δικαιώματος ε, της οικογενειακής ζωής και της ιδιωτικής σφαίρας. Ε, αυτό επίσης είναι ένας λόγος για να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και η Κομισιόν νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθεί προς κάπως διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που μας περιέγραψε. Η κυρία δεν θέλω να δημιουργήσω εχθρού, αλλά νομίζω ότι κάτι πρέπει να σημειώσουμε εδώ. Προερχόμενοι από ένα κόμμα που προσπαθούσε να υπερασπιστεί τις σχέσεις μεταξύ του ατόμων του ιδίου φίλου στη Δανία, που το 89 ήταν η πρώτη χώρα που θέσπισε κάτι σχετικό, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να επιβάλλουμε δια της βίας κάτι σε άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει να επιβάσουμε διατάξεις κατά της διακριτικής μεταχείρισης. Αυτό και βέβαια πρέπει να το κάνουμε. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα για το άρθρο 7. Όμως δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την άμβλωση στην Ιρλανδία, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στην Πολωνία την νομοθεσία αυτή, διότι η επικουρικότητα αναφέρεται σαφώς στη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτά αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία και σαφώς ε, συμφωνούμε με την ελεύθερη κυκλοφορία και εγώ είμαι υπέρ του να αποδεχθεί η Πολωνία αυτό που συζητάμε εδώ. Δεν νομίζω όμως ότι θα ήταν σκόπιμο να επιβάλλουμε κάτι χωρίς διάλογο. Τώρα στη Δανία με το πέρασμα των χρόνων έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα. Όμως καθ' όλη αυτή τη διάρκεια σεβόμαστε το φόβο των ανθρώπων και γι' αυτό θέλω και στο τωρινό θέμα να επισημάνω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχεις δίκιο, Μάικλ, ότι το κομμάτι που έχει σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία σε αυτό το θέμα είναι σαφές και δεν θα πρέπει να παραβιάζει την κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν μπορούμε όμως να επιβάλλουμε τη δική μας συγκεκριμένη νομοθεσία σε άλλες χώρες. Αυτή είναι η δική μου θέση, παρότι είμαι υπέρ όλων των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων. Ευχαριστώ την κυρία Όκεν. Θέλει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσθέσει κάτι. Δεν θέλω να ξανανοίξουμε τη συζήτηση. Πολύ σύντομα το κύριο μήνυμά μου δεν θέλω να χαθεί. Είναι θετικό. Θα εξετάσουμε την πρακτική που ισχύει στην Πολωνία από την οπτική γωνία της παραβής του κοινοτικού δικαίου και την επιπτώσεων που έχει τους κοινοτικού πολίτες όσον αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. Θέλουμε να γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώματα. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη όταν εμείς κάνουμε κοινοτική νομοθεσία. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε ακόμη μια φορά και θέλουμε όλες οι χώρες να σέβουν την κοινοτική νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος των αναφερόντων θέλει να απαντήσει. Του δίνω ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ και πάλι. Μα αφήσετε να παρουσιάσουμε το πρόβλημά μας. Νομίζω ότι πρέπει να εστιαστούμε στο κύριο πρόβλημα, που είναι το γεγονός ότι, και το είπε απολύτω σαφώ ο κύριος Κάσμαν, το θέμα είναι ότι οι Πολωνοί πολίτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα ε, κυκλοφορία σε άλλες χώρες και αλλοδαποί δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να ζήσουν μαζί με Πολωνούς πολίτες. Αυτό θα ήθελα να πω ώστε να γίνουν κάποιες προτάσεις για λεγές στο οικονομικό δίκαιο στην Πολωνία. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τις διάφορες παρεμβάσεις και φαίνεται με σαφήνεια ότι θα παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Αλλά εδώ πρέπει να πω ότι δεν έχουμε ειδικέ αρμοδιότητες. Εκτιμούμε το ανοιχτό πνεύμα με το οποίο αντιμετωπίζει η Κομισιόν το θέμα αυτό. Και θα πρέπει Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι αρμόδια περισσότερο από εμάς για αυτά τα θέματα να συνεχίσει να εξετάζει την κατάσταση. Είπε ότι θα δει η Κομισιόν κατά πόσον υπάρχει διακριτική μεταχείριση ή όχι στα πλαίσια της αναφοράς. Και όπως αναφέρθηκε, εμείς έχουμε κάποιες αρμοδιότητες, τα πλαίσια αυτών θα κινηθούμε, ούτως ή άλλως είμαστε τα οποιασδήποτε μορφής διάκρισης, όχι μόνο διότι έχουμε την σχετική οδηγία, αλλά διότι τα δικαιώματα του κάθε πολίτη θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και κανένας δεν θα πρέπει να μπαίνει στο περιθώριο για οποιαδήποτε επιλογή του. ακούσουμε τι μας είπε για αυτά τα θέματα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε ένα σημείωμα στις πολωνικές αρχές στο οποίο βεβαίως δεν μπορούμε να προτείνουμε να αλλάξει η δική τους νομοθεσία, το οποίο και αναφέρον, αλλά μπορούμε να τους πούμε ότι ε, η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβλήματα και όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και για άλλες παρεμφερείς και περιμένουμε να μας δώσουν κάποιες εξηγήσεις σε σχέση με αυτή την κατάσταση οι πολωνικές αρχές. Όλα αυτά στα πλαίσια της διακριτικής μεταχείρισης κάποιων πολιτών αλλά θα παραμείνει η αναφορά ανοιχτή, όπως είπαμε. Είναι ομόφωνη αυτή η απόφαση της Επιτροπής. Παραμένει η αναφορά αυτή ανοιχτή. Σας ευχαριστώ και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, την αναφορά 829-208 του κυρίου Φερνάντο Σουάρες η οποία εξετάστηκε από κοινού με την ε, αναφορά 1085. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Κούκεν, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, γιατί αναφέροντας δεν είναι παρόντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη δόθηκε ένα θετικό σήμα προς την Επιτροπή σας ε, στο παρελθόν, ε, λέγοντας ότι μετά τις δραστηριότητε μας προς τις γαλλικές αρχές, η γαλλική Βουλή τον Απρίλιο του 2009 άλλαξε τον αστικό κώδικα γιατί όπως γνωρίζετε αυτό ήταν ένα από τα βασικά εμπόδια στη Γαλλία. Ότι η Γαλλία δηλαδή δεν αναγνώριζε τα αστικά σύμφωνα συμβίωσης που είχαν συναυθεί σε άλλη χώρα και δεν τους έδινε την ίδια νομική ισχύ, ιδίως στα θέματα φορολογίας. Επενέβη λοιπόν η Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, αυτό δείχνει την δέσμευσή μας κατά της ομοφοβίας και την πρόθεσή μας να τηρείται η νομοθεσία κατά της διακριτικής μεταχείρισης από όλα τα κράτη-μέλη. Όσο έχει η κατάσταση τώρα στη Γαλλία και αυτό φαίνεται και από την τελευταία ανακοίνωση από τη Γαλλία που λάβαμε στις 3 Μαρτίου του 2010, όταν συνάπτει κανείς ε, ένα σύμφωνο συμβίωση στην Αγγλία, που ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση η υπόθεση του αναφέροντος ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος και ε, μετακομίζει κάποιος στη Γαλλία, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Οδηγίας για την Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Γαλλία τώρα έχει αλλάξει την νομοθεσία και χορηγεί τα ίδια πλεονεκτήματα και σε άλλους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μη Γάλλους, όπως και στους ε, Γάλλους ε, πολίτες που συνάπτουν το Γαλλικό Αστικό Σύμφωνο Αλληλεγγύης. Όσον αφορά την παρούσα αναφορά, υπάρχουν δύο συγκεκριμένες συνέπειες. για δύο καθήκοντα. Καταρχήν για το φόρο κληρονομίας και για την νομοθεσία που ισχύει για τις ε, ε, ε, δωρεές και μεταφορές περιουσίας εν ζωή, όπως επίσης και για το φόρο εισοδήματος δεν έλαβε περαιτέρω πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον αναφέροντα. Είχαμε έρθει σε επαφή με τον αναφέροντα στις 8 Ιουλίου του 2009 τελευταία φορά και του ζητήσαμε να υποβάλει πληροφορίες ε, για τις πρακτικές επιπτώσεις, για το αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση για τον αναφέροντα ή αν ε, υπάρχει κάποιο, υπάρχουν κάποιες άλλες δυσκολίες. Δεν έχουμε όμως λάβει απάντηση από τον αναφέροντα Υποθέτουμε λοιπόν ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον δυσκολίες ο αναφέρον ή έχει βελτιωθεί η κατάσταση για τον αναφέροντα και ότι τα μέτρα που έχει λάβει η Γαλλία είχαν τελικά θετικές συνέπειες για τα αστικά σύμφωνα συμβίωσης που συνάπτονται στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Ο κ. Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως είπα και προηγουμένως η δήλωση της ε, Αντιπροέδρου της Επιτροπής της κυρίας Ρέντινγκ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και φαίνεται ότι ε, κινούμαστε σε ένα σύστημα δύο ε, τροχιών, δηλαδή οι χώρες που έχουν αστικά σύμφωνα συμβίωση για άτομα του ίδιου φίλου. μπαίνουν σε ένα είδος αμοιβέ αναγνώρισης και υπάρχει και η άλλη ομάδα χωρών που ακόμη δεν προσφέρουν αυτά τα δικαιώματα σε ε, άτομα του ίδιου φίλου που θέλουν να συμβιώσουν. Είχαμε διαπραγματευτεί αυτό το θέμα και με την προηγούμενη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου και είχαμε ζητήσει να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Και νομίζω, χωρί να είμαι απολύτω βέβαιο, γιατί δεν είναι το κόμμα μου πλέον στην κυβέρνηση, πιστεύω ότι ε, γίνονται διαπραγματεύσει και με την Ισπανική κυβέρνηση για να διασφαλίσουμε την αμοιβαία αναγνώριση. Οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με άλλε χώρε, Βέλγιο, Ολλανδία κλπ. Προσπαθώντας να εξετάσουμε ένα μοντέλο βάσει του οποίου με μια απλή συμφωνία μια χώρα που έχει αστικά σύμφωνα συμβίωσης για άτομα του ιδίου φύλου μπορεί αν υπογράψει τη συμφωνία να δώσει αναγνώριση και στην άλλη χώρα χωρίς να χορηγεί υπερισχύοντα δικαιώματα. Απλώς αμοιβαία αναγνώριση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλή η τρέχουσα κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Θα μπορούσε να μείνει ανοιχτή η αναφορά όσο συνεχίζει τι εργασίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πιθανά μέτρα αμοιβέ αναγνώριση. Αλλά όπω είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή φαίνεται να έχει επιληθεί το πρόβλημα του συγκεκριμένου αναφέροντο, θα μπορούσε να κλείσει η αναφορά, αλλά θα σημειώσουμε στα πρακτικά ότι συνεχίζεται το θέμα σε άλλε χώρε. Ευχαριστώ. Grazie collega Cashman, non c'è nessun altro che intervenire. Ευχαριστώ. Θέλει κανένα συνάδελφο να λάβει το λόγο. Ακούσαμε τι είπε η συνάδελφη, ακούσαμε τι είπε και ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή, ο οποίο δήλωσε ότι αναφορά αυτή παρά το γεγονό ότι περιέχει ακόμη κάποια προβλήματα που υπάρχουν σε κάποιες χώρες, έχει σημειώσει μια κάποια πρόοδο, διότι υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα, παρά το γεγονός δεν μπορούμε να το πούμε με μαθηματική βίβλια. Ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι θα πρέπει να απευθυνθεί και πάλι ο αναφέρον στις γαλλικές αρχές για να δει κατά πόσον έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Αυτό ισχύει και για τις δύο αναφορές. Μετά από την δήλωση της Επιτροπής μπορώ να θεωρήσω ότι έχει ναι, ξεπεραστεί οι δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά θα ήθελα η Επιτροπή να μας το επιβεβαιώσει αυτό, δεδομένου ότι εξέφρασε κάποιες αμφιβολίες. αλλά φαντάζομαι ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει κλείσει ικανοποιητικά η αναφορά αυτή. Περνούμε στην επόμενη. 305 τη κυρία Μαρίζα Πινιόλο, Ιταλική Συνταγενιστικά είναι ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνω στην Κομισιό αμέσω το λόγο. Ναι, κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για μια πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλική καταγωγή που ζει στο Βέλγιο από τότε που γεννήθηκε. Η αναφορά αφορά το σύζυγό της που είναι από τη Σενεγάλη που μετά από το γάμο του με την αναφέρουσα συνέχισε να διαμένει στη Σενεγάλη. Το ζεύγος απευθύνθηκε στην Σενεγάλη, στη Βελγική Πρεσβεία για να πάρει θεώρηση όπως προβλέπεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 της σχετικής οδηγίας 38-2009. Του αρνήθηκαν τη θεώρηση και του κοινοποιήθηκε η απόφαση στις 8 Ιουλίου 2008 διότι όπως ελέγχθη δεν υπήρχε απόδειξη του οικογενειακού δεσμού. Φαίνεται ότι ο γάμος έγινε στις 4 Απριλίου 2008 μεταξύ της Ιταλίδας και του Σενεγαλέζου αλλά το πιστοποιητικό ε, γάμου δεν κατοχυρώθηκε και στο Βέλγιο. Έχετε ούτως ή άλλως αντιγραφή του πιστοποιητικού γάμου και δεν ίσως αναφέρεται ότι ήταν ήδη χωρισμένη η αναφέρουσα. Οι Βέλγοι υπάλληλοι λοιπόν έφτασαν στο αποτέλεσμα ότι δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αυτός ο οικογενειακός δεσμός. Εφεσίβαλε ε, κατά της απόφασης αυτής τον λόγο ζεύγος, απερίφθη η έφεση, διότι σύμφωνα με τους Βέλγους η έφεση υπευλήθη καθυστερημένα. Δηλαδή, ε, πέραν των τα την κοινοποίηση της άρνης χορήγης θεωρίας. Ο σύζυγος απευθύνθηκε στην ε, Ιταλική, στο Ιταλικό προξενείο και έλαβε μία θεώρηση τύπου Δέλτα. Αλφαβήτα γάμα Δέλτα. Δεδομένου ότι η σύζυγός του είχε την Ιταλική επικότητα. Και μετά υπέβαλε αίτηση για οικογενειακή επανένωση στις βελγικές ε, αρχές της 6 Τετάρτου του 2010. Μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρακολουθεί την όλη υπόθεση χάρη στην ε, κοινοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε εξηγήσει ε, στους εκπροσώπους της βελγικής κυβέρνησης και του υπεύθυνου Υπουργείου και ο Σενεγαλέζος σύζυγος της αναφέρουσας, στις 20 Σεπτεμβρίου του 2010, πήρε άδεια παραμονή στο Βέλγιο. Ως μέλος οικογένειας ε, κοινοτικού πολίτη στα πλαίσια της σχετικής οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 313 του 2009 σε θέματα γενικών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά αφορά τα δικαιώματα διαμονής και εισόδου στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατήρησε ότι τα μέλη της οικογένειας που δεν έχουν κοινοτική επικότητα όχι μόνο έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στην κοινοτική επικνάτεια αλλά και να τύχουν θεώρησης εισόδου. Αυτό σύμφωνα με τα ανακοίνωση που κάναμε το 2009. Και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε 503 κάθετος 2003. Απόφαση κατά της Ισπανίας. Εκεί αναφέρονται από το δικαστήριο ποια είναι τα δικαιώματα των κοινωνικών πολιτών. Και αυτή ήταν η διαφορά, όπως είπαμε, στην ε, ανακοίνωση του 2009 μεταξύ μελών μιας οικογένειας και, τρίτο, και επικών τρίτων χρόνων που δεν έχουν οικογενειακούς δεσμούς. Συμπερασματικά, όσον αφορά το δικαίωμα που έχει ο σύζυγος να αποκτήσει θεώρηση εισόδου, στην ανακοίνωση του 2009 με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνεμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς ενημέρωση, αλλά κυρίως στα κράτη-μέλη που πρέπει να εφαρμόσουν το κοινοτικό δίκαιο, Αναφέρουμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να απαιτήσουν μόνο την παρουσίαση ενός ε, έγκυρου διαβατηρίου και την απόδειξη ότι υπάρχει οικογενειακός δεσμός με τον κοινοτικό πολίτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Σενεγαλέζος κύριος μπορεί να αποδείξει ότι έχει νυμφευθεί την ε, αναφέρουσα, την Ιταλίδα. Κανένα συμπληρωματικό έγγραφο δεν μπορεί να ζητηθεί καμία άλλη απόδειξη ότι κάποιος τον έχει προσκαλέσει κτλ. Παρά το γεγονός ότι λύθηκε αυτή η προσωπική, το προσωπικό πρόβλημα του κυρίου αυτού με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζουμε τη βελγική νομοθεσία όσον αφορά τη χορήγηση θεώρησης σε μη κοινοτικούς συζύγους κοινοτικών πολιτών και επιφυλάσσουμε την συνέχεια που θα δώσουμε στην υπόθεση αυτή βάση της εξέτασης αυτής. Εάν οι αξιότιμοι βουλευτές συμφωνούν, προτείνουμε να κλείσει αυτή η αναφορά, δεδομένου ότι το πρόβλημα λύθηκε για τον Σενεγαλέζο κύριο. Ευχαριστώ. Υποθέτω ότι συμφωνούμε όλοι, δεν υπάρχει αντίρρηση, ας κλείσει αυτή η αναφορά. Να κλείσει λοιπόν αυτή η αναφορά. Συμφώνουμε όλοι, λέει η πρόεδρο. Και ευχαριστούμε την Κομισιό για αυτή την εμπεριστατωμένη εξήγηση που μας έδωσε. Περνάμε στο επόμενο θέμα 21. 1837 Παύλα 2009 του Ρομπέρτο Μαρκότσο. Και πάλι δίδε το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, Τόμας Ντόνκβιστ. Ε, ευχαριστώ. Σε αυτή την αναφορά ο κύριος Μαρκότσο, Ιταλικής Ιθαγένειας, αναφέρει ότι στην απόφαση να... Σύμφωνα με την απόφαση 2009-1837 σχετικά με... και την νομοθεσία πλαίσιο, θα πρέπει να γίνεται ένα βιντεοσκόπηση των ανακρίσεων της αστυνομίας. Και θα πρέπει ε, να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων σε ποινικέ αποθέσει και μεταφορά κατά δίκον. Αυτό ε, είναι ε, θέμα προστασίας των δικαιωμάτων των υπηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου περί αποφάσεων που κοινοποιούνται σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται όταν επιβάλλονται ποινές ε, που έχουν επιβληθεί από άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστροφα. Το συμπέρασμα της Κομισιόν είναι ότι συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι χρειάζεται μηχανισμός που θα διασφαλίζει ότι δικαιώματα στις ποινικέ διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατεύονται και η Κομισιόν αποπειράθηκε ήδη μία φορά πριν να προτείνει νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή των διαδικασιών. Αλλά όμως ε, η προσπάθεια αυτή δεν καρποφόρησε. εξαιτίας των θέσεων των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την πρόταση αυτή ως μέρος μεγαλύτερης εξέτασης των δικονομικών δικαιωμάτων που αφορούν την ε, απονομή της δικαιοσύνης, αλλά θα χρειαστούν κάποια χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του οδικού χάρτη το 2014 το νωρίτερο. Αυτό εν συντομία, αυτή εν συντομία είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Παρεμβάσεις παρακαλώ, ο κύριος Μπουσινά. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον αναφέροντα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις καταχρηστικών πρακτικών κατά την ανακριτική διαδικασία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταχρηστικές πρακτικές που σε τελευταία ανάλυση άπτονται θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, νομικών διαδικασιών κλπ. Αν υπάρχει καταγραφή, αυτό θα είναι ένα ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο για την προάσπιση δικαιωμάτων σε ένα εφετείο σε οποιαδήποτε υπόθεση και συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του αναφέροντος. Και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει αυτή την περίοδο βραχύνοντας ε, τη διάρκεια αναμονής όχι να περιμένουμε κάποια χρόνια όπως είπατε, θα πρέπει να είναι το διάστημα αυτό όσο γίνεται βραχύτερο, γιατί είναι ζωτική σημασία σε πολλές χώρες και στη δική μου επίσης, στη Ρουμανία. Γιατί παραβιάζονται βασικοί κανόνες ε, και η παραβίαση αυτή είναι απαράδεκτη. δεν υπάρχουν εμπόδια, ούτε τεχνικά ούτε οικονομικά, για να μην εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει σύντομα με μια έκθεση πρόοδου για την εφαρμογή της ε, διαδικασίας καταγραφής ε, των ανακρίσεων. Ευχαριστώ κύριε Μποσινάρο. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς κατά. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ βέβαια με όσα ακούσαμε. Λέτε ότι κάποια κράτη-μέλη αρνούνται ε, το σύστημα των δικαστηρίων ακολούθησε τη διαδικασία εναρμόνισης. Τα κράτη-μέλη ήθελαν να κρατήσουν το δικαστικό σύστημα σε εθνικό επίπεδο. Κατανοητός συντηρητισμός. Θα ήθελα όμως να μου πείτε τι επιχειρήματα προβλήθηκαν, γιατί εδώ δεν πρόκειται για το σύστημα των εθνικών δικαστηρίων. Αν υπάρχει ένα κοινό σύστημα, πώς θα ξέρουμε τι έχει γίνει όταν δεχόμαστε ετοιμιγορίες δικαστηρίων άλλων χωρών. Θα με ενδιέφερε να ξέρω ποια ήταν τα επιχειρήματα για την απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή τι είπανε, να μην ανακατεύεστε στα, στις εσωτερικές μας υποθέσεις ή υπήρξαν σοβαρά επιχειρήματα που θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Συμφωνώ να μείνει ανοιχτή η αναφορά, αλλά είμαι περίεργη για τον όλο χειρισμό και την πορεία που ακολούθησε το θέμα. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απαντήσει. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν είναι δική μου υπόθεση και φάκελος. Δεν γνωρίζω τι επιχειρήματα προέβαλαν τα κράτη-μέλη. Μπορώ όμως να μάθω και να σας ενημερώσω. Να ενημερώσω την Επιτροπή σας δηλαδή, αν θέλετε. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει ακόμα να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Λάβαμε υπόψη μας τις διευκρινήσεις του εκπροσώπου της Επιτροπής. και ελπίζομαι ότι και πριν από το 2014 θα δώσει κάποια καινούργια στοιχεία προόδου η Κομισιόν μετά από πρόταση της γραμματείας θα έλεγα ότι πρέπει να στείλουμε ένα σημείωμα και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που ασχολείται επίσης με το ζήτημα αυτό. Έτσι θα μπορούμε να ε, συνεννοηθούμε και με τις άλλες αρμόδιες επιτροπές. Παραμένει ανοιχτή αναφορά. Τώρα. Στις 16.30 ε, θα έρθει η Επίτροπος Ρέντινγκ. Τελειώσαμε λίγο νωρίτερα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στις άλλες αναφορές, οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα. Colleghi, riprendiamo i lavori. Επανέλθουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε μαζί μα την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω εξ ονόματο τη Επιτροπή μου για την παρουσία τη. Είναι η δεύτερη φορά που μα τιμά με την παρουσία. Σήμερα το απόγευμα η κυρία Επίτροπος θα μας παρουσιάσει την τελευταία έκθεσή της για την Ιθαγένεια που παρουσίασε πρόσφατα και είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας. Η Επίτροπος θα πρέπει να μας αφήσει σε μία ώρα και της δίνω χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση το λόγο και μετά θα δούμε πώς θα οργανώσουμε στο τέλος της παρέμβασης κυρίας Επιτρόπου τις ερωτήσεις. Κυρία Πρόεδρε. Μου, μου θυμίζετε παλιές εποχές. Ιταλική Προεδρία, Ιταλή Πρόεδρος. Και εγώ έφυγα εδώ και 20 χρόνια από εδώ και μετά από μένα ήταν Ιταλίδα η Πρόεδρος. Καταρχάς εγώ ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής αυτής και μετά έγινε η Ρόζα Μπίντι, Ιταλίδα. Κυρία Πρόεδρε, σωστά είπατε ότι θα σας μιλήσω για την νέα έκθεση που αφορά την Ιθαγένεια και παρουσιάστηκε στις 27 Οκτωβρίου, όπως ξέρετε. Αυτό ακολουθεί τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2009 ο πρόεδρος και είπε με σαφήνεια ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει ανθρωποκεντρική πολιτική κυρίως και για να υπογραμμίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για τους πολίτες και για να άρουμε όλα τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμη στην ενιαία εσωτερική αγορά, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως για τους πολίτες. Επίσης, μάθαμε πολλά από την έκθεση Ντολαμασούρ του 2008, την οποία είχε συντάξει ο συνάδελφός σας, ο κύριος Ντολαμασούρ και ο οποίο απαρίθμησε με συγκεκριμένο τρόπο τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτε στην καθημερινή του ζωή αν θέλουν να υποφεληθούν από την ενιαία εσωτερική αγορά. Εμπνευστήκαμε λοιπόν πάρα πολύ από την έκθεση και εκ τώρα εγώ συνέταξα την έκθεσή μου αυτή για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια που είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται από Επίτροπη που ασχολείται με όλα τα καθημερινά πρακτικά προβλήματα των πολιτών που είναι εργαζόμενοι, ταξιδιώτες, φοιτητές που θέλουν να παντρευτούν, να αγοράσουν μια διεκτησία, να τύχουν ιατρικής περίθαλψης, οτιδήποτε μπορούν να κάνουν στην καθημερινή του ζωή. Παρουσίασα εγώ 25 σύντομες δράσεις, βράχοι και μεσοπρόθεσμες. Και νομίζω ότι θα λάβετε κάποια σχετικά έγγραφα όπου κυρίως αναφέρονται τα κύρια θέματα πραγματεύουμε στην έκθεσή μου. Κυρίως αναφέρομαι στους πολίτες που ζουν σε ένα άλλο κράτος μέλος και πρέπει να χαίρουν του δικαιώματος ελεύθερης διαμονής και διακίνησης. Πρόκειται εδώ τουλάχιστον για 12 εκατομμύρια άτομα τα οποία ζουν. Και σε ερωτήσεις που έγιναν, πάρα πολλά εκατομμύρια είπαν ότι θα ήθελαν να μπορούν να μετακινούνται, αλλά πιστεύουν ότι είναι πολύ πλοκό και δεν το κάνουν αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει εμπόδιο. Δεν θα υποχρεώσουμε κανένα να κάνει τίποτα, αλλά εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να άρουμε τα εμπόδια και όταν κάποιος αποφασίσει να μετακινηθεί, να πάει σε άλλη χώρα... Μπορεί... Επίσης, υποβάλαμε ερωτήσει αυτού οι οποίοι μετακινήθηκαν και είμαστε ότι τουλάχιστον οι μισοί αντιμετώπισαν δυσκολίε και διοικητικέ καθυστερήσει. Εκτό από τα καθημερινά προβλήματα, Λοιπόν, προστίθενται και αυτά τα διοικητικά. Οι διοικητικέ δυσκολίες οι οποίες προστίθενται σε όλα τα άλλα προβλήματα που πρέπει ο καθένας να αντιμετωπίσει στη χώρα του. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα ώστε να είμαστε και σίγουροι ότι εφαρμόζονται σωστά οι κοινοτικοί κανόνες από τα κράτη-μέλη. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δεν είναι τι θα κάνουμε με τους νέους νόμους, αλλά εάν εφαρμόζονται και ισχύουν σωστά οι κανόνες που ισχύουν. Εάν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Εάν υπάρχει η ίδια μεταχείριση σε διοικητικό επίπεδο. Εάν όλοι οι φορεί σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο σε κάθε κράτο γνωρίζουν την κοινοτική νομοθεσία, διότι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μόνο κακοπιστή αλλά και άγνοια των κοινοτική νομοθεσία. Και κάτι που μου φαίνεται επίση σημαντικό είναι ότι και οι ίδιοι οι πολίτε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά του. Πορεία από αυτοί δεν τα γνωρίζουν. Ένα τρίτον των πολιτών μα λέγουν αμέσω ότι δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν ποια ήταν τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση λοιπόν αυτή αναφέρουμε και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ε, ε, πολίτες που ζουν σε μια άλλη χώρα για τα ε, εκλογικά τους δικαιώματα. Και εδώ υπάρχει έλλειψη γνώσεων, αλλά υπάρχουν και κάποια σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την ε, καταχώρηση πολιτών σε ε, εκλογικού καταλόγους μιας άλλης χώρας. Γι' αυτό χρειάζονται να έχουν μια ταυτότητα. Και ποιοι είναι οι περιορισμοί που υφίστανται εάν θέλουν να ψηφίσουν για ένα πολιτικό κόμμα ή να ε, προσχωρήσουν σε ένα πολιτικό κόμμα, να εκλεγούν σύμφωνα με ένα άλλο κόμμα. Έγιναν διάφορες έρευνες το 2010 που αποδεικνύουν και ήδη το είπα ότι λιγότερο από ένα Τρίτον, 32% των πολιτών θεωρούν ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους. 70% των Ευρωπαίων δηλαδή δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν δίκτυα κοινοτικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση προβλημάτων. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ε, τα δίκτυα, το δίκτυο Solvit για την επίλυση των προβλημάτων, αλλά πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες. Εάν δεν το γνωρίζουν, δεν τα χρησιμοποιούν. Άρα δεν είναι αποδοτικά αυτά τα δίκτυα. Δεδομένου ότι τα πράγματα είναι τόσο πολύπλοκα και δεδομένου ότι υπάρχουν τόσο πολλά δίκτυα, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να κάνει αυτό που λέγεται one-stop shop μία ιστοσελίδα που λέγεται Your Europe, η Ευρώπη σας, όπου θα μπορούν οι πολίτες να κάνουν ερωτήσεις, να υποβάλουν ερωτήσεις και θα κατευθύνεται αυτομάτως αυτόν ο οποίος θα του δώσει την κατάλληλη απάντηση. Δεν θα ξέρει τι γίνεται πίσω από την οθόνη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το χρειάζεται κιόλα. Αυτό που χρειάζεται είναι να ξέρει ότι σε αυτή την ιστοσελίδα θα απευθύνω την ερώτησή μου και θα πάρω την σωστή απάντηση και θα βοηθηθώ. Αυτό βεβαίως γίνεται συνεργαστή με το Europe Direct που γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσά πολύ καλά. Uh, have Τελικά μπορούν να κάνουν το παράπονά τους οι πολίτες Ευρωπαίοι σε εσά εδώ στην Επιτροπή Αναφορών που είναι πάρα πολύ σημαντική και σε, αυτή την, ε, σε αυτόν τον ιστότοπο όπου απευθείας μπορούν ε, να υποβάλουν ερωτήσεις και να κάνουν τα παραπονά τους οι αναφορές. Σιγά σιγά λοιπόν γίνεται όλο και πιο σημαντικό από το διάστημα. Πριν από το τέλος του 2010 εγκρίναμε την ε, στρατηγική αναπηρία στα πλαίσια της στρατηγικής 12-20 ε, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, αναπήρων. Έχουμε Επίσης, δες και ε, κίνηση την ε, πράσινη βίβλο για τη μείωση της γραφειοκρατίας και για να διευκολύνουμε τη ζωή των πολιτών. Όταν χρειάζεται να έχουν στην χώρα στην οποία διανέμουν ένα έγγραφο, ένα πιστοποιητικό από τη χώρα καταγωγής τους. Ε, Επίσης, ε, αυτή τη συμφωνία αστικής, οι συμφωνίες αστικής συμβίωσης είναι κάτι άλλο το οποίο μας ενδιαφέρει και θέλουμε να διευκολύνουμε και τις ε, διαδικασίες για να ξέρει κανείς αν θέλει να χωρίσει ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο. Τώρα προσπαθούμε επίσης τα θέματα της ε, χωρισμού της περιουσίας σε περίπτωση χωρισμού να τα επιλύσουμε. Θέματα τα οποία αφορούν ε, την προστασία κάποιων θυμάτων. Πολλές φορές κατά την διάρκεια ε, της ε, επαφής τους με τα δικαστήρια πολλά θύματα δεν λαμβάνονται στα σοβαρά και γίνονται θύματα στην επαφή τους κατά τη διάρκεια όλων των ε, διαδικασιών με τα δικαστήρια ή γίνονται για δεύτερη φορά θύματα. Όλα λοιπόν αυτά τα δικαιώματα προσπαθούμε να τα λάβουμε υπόψη. Στο ποινικό δίκαιο, όπως ξέρετε, υπάρχουν πάντα και τα δικαιώματα των ε, κατηγορουμένων να έχουν τη διερμηνία στη μετρική τους γλώσσα κατά τη διάρκεια της ακροματικής δικασίας. Ε, υπάρχει το δικαίωμα της ενημέρωσης και Εφέτος θεσπίζουμε και το δικαίωμα επικοινωνία με την οικογένεια και το δικαίωμα να τύχει τη βοήθεια ενό δικηγόρου ένα κατηγορούμενο. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία προετοιμάζουμε για φέτο, και αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς εδώ ψηφίζει για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη σχετική οδηγία και τα δικαιώματά τους Επίσης θα σας μιλήσω για το πακέτο μέτρων για τα ταξίδια που θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές και για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις νέες ανάγκες των καταναλωτών, στα πακέτα online που μπορεί, διακοπών που μπορεί ένας ε, πολίτης που θέλει να ταξιδέψει να ζητήσει και βεβαίως και τα δικαιώματα δικαστικής συνδρομής και συμβουλών που μπορεί να έχει κάποιος κοινωτικός πολίτης σε τρίτη χώρα. Όλα, όλα αυτά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους πολίτες μας. Έχουμε ξεκινήσει μία συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους οργανισμούς ε, και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία και να εντοπίσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να εμπλακούν και τα εθνικά κοινοβούλια στη συζήτηση αυτή. Όπως και εσείς, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Επιτροπή Αναφορών δίνεται τη δυνατότητα στους πολίτες να απευθυνθούν άμεσα σε εσά. Έτσι και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στους εθνικούς βουλευτές και η συγκέντρωση των ε, καταγγελιών των πολιτών θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει και τι περιμένουν οι πολίτες από μας. Όπως είπα και στην αρχή, Τελικά αυτό που θέλουμε δεν είναι απλώς η θέσπιση νέων ε, οδηγιών ή νέων κανονισμών. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το να γνωρίζουν οι πολίτες ότι έχουν αυτά τα δικαιώματα που έχουν. Και γι' αυτό το λόγο θα προτείνω στο Κολέγιο των Επιτρόπων, το, στο Κολέγιο των Επιτρόπων να είναι το 2013 να οριστεί ως ε, Ευρωπαϊκό Έτος για τους Ευρωπαίους πολίτες. Το 2013 θα έχουμε την 20η επέτειο της έσπισης της ε, Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας από την συνθήκη του Μάστριχ θα είναι και ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και θα είναι μια κατάλληλη χρονική στιγμή για να απευθυνθούμε στους πολίτες και να τους εξηγήσουμε ότι να, αυτά κάνει η Ευρώπη για να μπορείτε εσείς να αισθάνεστε περισσότερο ελεύθεροι και να αισθάνεστε ότι ε, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά σας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βελτιώσουμε λοιπόν την ε, γνώση των πολιτών για τα δικαιώματά τους και θα τους ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ισχυρή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως επίσης και με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα πιο ισχυρό μήνυμα. Το 2013, βάσει των προγραμμάτων μας, θα έχουμε επιλύσει πάρα πολλά προβλήματα και φραγμούς τους οποίους αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην εσωτερική αγορά. Θα έχουμε ε, την διαδικτυακή πύλη της μιας και μόνης θηρίδας, του One Stop Shop. Θα έχουμε λοιπόν ένα μήνυμα το οποίο μπορούμε να απευθύνουμε προς τους πολίτες και ένα σήμα το οποίο μπορούμε να τους δώσουμε για την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο ότι τα συμπεράσματα της δικής σας έκθεσης από τον Ιούνιο του 2010 συμπίπτουν με τα ευρήματα της έκθεσης ε, για την Ιθαγένεια διότι εντοπίζουν τα ίδια εμπόδια τα οποία εντοπίσαμε κι εμείς. Η έκθεσή σας είναι πολύ χρήσιμη, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε ποια είναι τα σημεία ε, στα οποία οι πολίτες της Ευρώπης νιώθουν ότι μπορούν, έχουν το δικαίωμα να σας στείλουν μια αναφορά, να σας στείλουν μια επιστολή ποια είναι τα σημεία στα οποία θεωρούν ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η Επιτροπή σας λοιπόν είναι πολύτιμος εταίρος για μας και γι' αυτό προσβλέπουμε και σε στενή συνεργασία και επικοδομητικό διάλογο σχετικά με τις προτεραιότητές μας και σχετικά με τα εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου επιτρέψατε να παρουσιάσω την έκθεση για την Ιθαγένεια και σας ευχαριστώ όλους που βοηθάτε να υλοποιηθεί και θα βοηθήσετε και κατά τα προσεχή έτη. Εάν συμφωνήσει το Κολέγιο των Επιτρόπων για την ανακήρυξη του 2013 ως έτους των πολιτών θα είναι κάτι στο οποίο θα εναποθέσουμε πολλές ελπίδες. Και το 2013 θα είναι έτος των πολιτών της Ευρώπης και το 2012 θα είναι ένα έτος προετοιμασίας για να μπορούμε το 2013 να θεσπίσουμε πολλές νέες πρωτοβουλίες και να είναι αυτό το έτος σημαντικό για ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Επιτροπό, την κυρία Ρέντινγκ. Η Επιτροπή μας σίγουρα θα υποστηρίξει την έκθεση αυτή και έχοντας ακούσει και αυτά που μας είπε η Επίτροπος κατανοούμε το εύρος των εργασιών σας και την ανάγκη συνεργασίας. Όλα τα εμπόδια τα οποία επισημαίνονται στην έκθεση μπορούν να συσχετιστούν με πολλές αναφορές τις οποίες εμείς λαμβάνουμε στην Επιτροπή μας. Είναι παρόμοια τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε και εμείς στην Επιτροπή μας. Και σήμερα εξετάσαμε διάφορα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την έκθεση αυτή. Σίγουρα λοιπόν θα ακολουθήσει επικοδομητική συνεργασία και τώρα ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι για το θέμα και θα δώσω κατευθείαν στην κυρία Βόλς το λόγο. Thank you very Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για την παρουσίαση. Για πολλούς από εμά που για κάποια χρόνια δραστηριοποιηθήκαμε στον τομέα της ηθαγένειας και των δικαιωμάτων στον τομέα αυτό, σας συγχαίρομαι για τις πολλές πρωτοβουλίες Υπάρχει ένα θέμα που, με το οποίο καταπιάνεται ο κύριος Λαμασούρ στην έκθεσή του για τα δικαιώματα, εκεί όπου ήδη υπάρχει νομοθεσία αλλά μπορούμε να την βελτιώσουμε και να την εφαρμόσουμε καλύτερα. Και είναι θαυμάσιο ότι θέλετε να αναδείξετε και ένα έτος. Πάντα έλεγα ότι χρειάζεται ε, μία όθηση για τα θέματα αυτά ε, όπως το 1992 και να μην αφήσουμε τα θέματα αυτά ε, χωρίς παρεμβάσεις. Πολλές εξαιρετικές ιδέες προβάλατε. Υπάρχει και ένα μέσο όπου πιστεύουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Ένα προβληματικό θέμα που το βλέπω και από τον αριθμό των email που δέχομαι είναι οι περιπτώσεις όπου ε, αποφάσισαν να ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας είτε για διαμονή ε, αποκλειστική σε μια άλλη χώρα είτε με διαλύματα και εκεί κάνουν μια μεγάλη αγορά. Αγοράζουν δηλαδή ένα κίνητο σε μια άλλη χώρα και τους προσφέρουμε προστασία ως καταναλωτές όταν αγοράζουν ηλεκτρονικά αγαθά τι προστασία όμως τους προσφέρουμε όταν κάνουν μια τόσο σοβαρή, ίσως τη μεγαλύτερη αγορά της ζωής τους σε μια άλλη χώρα μέλος. Είναι δύσκολο αυτό το θέμα γιατί άπτεται στο ευαίσθητο θέμα της εθνικής νομοθεσίας, αλλά σε περίπτωση διαζυγίου υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει και η συνήθις περίπτωση των πολιτών που κάνουν τέτοιου είδους αγορές. Και θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ δέχομαι email και άλλοι συνάδελφοι σίγουρα που συνδέονται με προβλήματα σχετικά με την αγορά γης ή ε, κατοικιών σε άλλη χώρα μέλος. Και αυτά τα θέματα υπάρχουν και στην Ισπανία, το ξέρετε, και αλλού. Δεν επιμένω σε αυτά. Τονίζω όμως ότι υπάρχει εδώ μια αναντιστοιχία η οποία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όσο εντείνεται η ελεύθερη κυκλοφορία. Γιατί γνωρίζουν τα βασικά δικαιώματα, το δικαίωμα ιδιοκτησίας που, που υπάρχει και στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι η θεωρία, ενώ η πρακτική είναι διαφορετική όταν προχωρούν σε αγορές σε άλλο κράτος μέλος. Το δικαίωμα είναι θεωρητικό, αλλά στην πράξη είναι συνειφασμένο με πολλές δυσκολίες. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και δύσκολο το θέμα αυτό και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, διότι το πρόβλημα συνεχίζεται και ε, πλήττει πολλούς πολίτες σε πολλές χώρες μέλη. Ευχαριστώ, η κυρία Στανόκα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και την αξιότιμη Επίτροπο για όλες τις πρωτοβουλίες της και είναι μεγάλη πρωτοβουλία αυτή να θεσμοθετηθεί ένα έτος ηθαγένειας. Όπως γνωρίζουμε όλοι, τώρα η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι άμεσο παράγωγο της ε, εθνικής ηθαγένειας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μόνιμα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται σε, στη, στη δικαιοδοσία κάποιων κρατών μελών, χωρίς όμως να έχουν την ηθαγένεια αυτού του κράτους μέλους. Αλλά δεν είναι και άλλο δαπή. Γιατί δεν έχουν ηθαγένεια άλλου κράτους. Αυτή είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που προβλέπεται από την νομοθεσία σε δύο βαλτικά κράτη, Λετωνία, Εσθονία και υπάρχουν μερικές εκατοντάδες πρόσωπα χωρίς ηθαγένεια. Είναι... Ζουν και στη Σλοβενία μερικοί ανηθαγενείς ή απροσδιόριστης ηθαγένειας άνθρωποι. Αυτό το πρόβλημα προέκυψε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της ε, Ιουγκοσλαβίας. Αυτά τα πρόσωπα λοιπόν υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους και έχουν ένα ειδικό καθεστώς στη Λετωνία και την Εστονία για παράδειγμα. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν ελεύθερα στη χώρα τους και έχουν και προξενική προστασία όταν είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή την προξενική προστασία του κράτους μέλους. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προτέρα νομοθεσία και με την επικούρηση των συναδέλφων, τον Μάικλ Κάσμαν και άλλους, μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε αυτή την κατηγορία των προσώπων και στις ρυθμίσεις για τις θεωρήσεις Επίσης ε, εντάσσονται μεταξύ εκείνων που έχουν ελεύθερο καθεστώς θεωρήσεων ε, στα μέλη της συνθήκης, με την εξαίρεση Βρετανίας και Ιρλανδίας, αλλά η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ισλανδία είναι χώρες που συμπεριλαμβάνονται. Είναι η Συμφωνία για την, ε, το ελεύθερο καθεστώς χορηγήσεων. Δεν πιστεύετε ότι μπορεί να διευρυνθεί η έννοια της ευρωπαϊκής ηθαγένειας ώστε να συμπεριλάβει και αυτά τα πρόσωπα που έχουν αυτό το ειδικό καθεστώς. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Εδώ στην Επιτροπή Αναφορών εξετάσαμε έναν αριθμό αναφορών από, από ανιθαγενείς από τη Λετωνία στη, που ζητούσαν την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τους χορηγηθούν δικαιώματα συμμετοχής στις εκλογές, γιατί δεν μπορούν να συμμετέχουν σε εκλογές καθόλου. Αυτή η υπόθεση έγινε ιδιαίτερη, γιατί με την, τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν όλοι οι, πίκο, οι ε, κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν. Αυτή όμως όχι. Και επειδή υπάρχει και μία αναφορά από την Εστονία που αναφέρεται στο δικαίωμα του εκλέγην στις ευρωπαϊκές εκλογές, ερωτώ. Δεν πιστεύετε ότι χρειάζεται ίσως ένας καινούριος κανονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ρυθμίζει το ποιος έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε τοπικές εκλογές, δημοτικές εκλογές και ευρωπαϊκές εκλογές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλα όσα είπε η κυρία Στανόκα, ιδιαίτερα σε εκείνους που θεωρούνται ανιθαγενείς και που είναι περίπου μισό εκατομμύριο τώρα. Κυρία Επίτροπε, δεν αμφισβητώ ότι είστε απόλυτα αφοσιωμένοι στο θέμα της ηθαγένειας, τα ίσα δικαιώματα. Αυτό το είπαμε και το διαπιστώσαμε πολλές φορές και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Υπάρχει όμως φαίνεται μια στενή ερμηνεία και νομίζω ότι υπάρχει, επειδή γίνεται μάχη, υπάρχει στενή ερμηνεία του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και γι' αυτό θεωρείται ότι υπάρχει ένα κενό γιατί ε, αφορά τον, ε, την ε, κοινοτική νομοθεσία, αλλά υπάρχουν και, υπάρχουν και εσωτερικά δίκαια τα οποία είναι σε αντίφαση. Εσείς ε, σίγουρα θέλετε να ασχοληθείτε με το θέμα στην Επιτροπή, αλλά από τα κράτη-μέλη υπάρχει κάποια προθυμία. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Είστε διατεθειμένοι να πιστείτε και ξέρω ότι πάντα, κυρία Αντιπρόεδρε και Επίτροπε, είστε ανοιχτοί να τροποποιήσετε το χάρτη ούτως ώστε να αποκτήσει νόημα το κείμενο αυτό και να μπορεί να παρατίθεται όταν πρόκειται για παραβιάσεις ε, του δικαίου ιδιοκτησίας, του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Αναφέρομαι στο άρθρο 17 ειδικότερα, γιατί υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα που τα βλέπουμε εδώ. Μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή, το έτος Ευρωπαϊκής Θεγένειας 2013. Εμείς ε, ασχολούμεθα με τα προβλήματα Ευρωπαίων πολιτών που θεωρούν ότι δεν έχουν ίσα δικαιώματα. Ε, ας πούμε το θέμα των, των οικοπεδοφάγων στην Ισπανία η αγορά παράνομων όμως ε, ακινήτων ε, και το θέμα της προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας θα πρέπει σε ολόκληρη την Ένωση να τύχει προστασίας. Επίσης ακούσαμε σήμερα ότι για όλο αυτό το θέμα της μη αναγνώρισης των ελεύθερων συμβιώσεων κλπ. Σήμερα από την Πολωνία είχαμε ένα περιστατικό όπου όταν υπάρχει τέτοια σύναψη καταχωρισμένη συμβίωση σε άλλη χώρα μέλος, εκεί από τη χώρα προέλευσής τους δεν ε, αναγνωρίζεται η σχέση αυτή είστε διατεθειμένοι να κάνετε μια μελέτη για λογαριασμό της Κομισιόν. Είναι κατεπήγον για να επανεξετάσετε την νομοθεσία στα κράτη-μέλη όταν αντιβαίνει στη Συμφωνία της Λισαβόνας και στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων ώστε να αρχίσει μια συζήτηση για το πώς θα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν αυτό το σημαντικό θέμα της σύγκρουσης με τον σημαντικό χάρτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την πολύ καλή έκθεση και για τα στοιχεία που μας δίνει σχετικά με τους Ευρωπαίους πολίτες. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θέτουμε στο επίκεντρο των προσπαθειών μας ε, την επίγνωση των πολιτών. Ο κ. Κάσμαν διορθώνει. μου αρέσουν τα πολωνικά, αλλά δεν τα καταλαβαίνω εγώ που είμαι Άγγλος μεταφράζονται στα πολωνικά αυτά που ακούω και όχι στα αγγλικά ε, και γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω τη διερμηνία. Μάλλον έκανα λάθος στα ακουστικά όμως ο κύριος Κάσμα. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Είχα πάρει λάθος ακουστικά. Βλέπετε, οι πολιτικοί συχνά έχουν ιδέες, αλλά ο εγκέφαλός τους ε, απορρίπτει τις ιδέες. Έχω μια ερώτηση σχετικά με το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούμε όταν λέμε ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας εντάσσεται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα από το Ραμπόρια Μπράβα, μια μικρή πόλη στην Ισπανία, όπου οι εκπρόσωποι των πολιτών μου έστειλαν ε, ε, μια επιστολή ε, και η ερμηνεία που ε, έχει δοθεί είναι ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής το θέμα που τους απασχολεί. Θα ήθελα να έχω μια απάντηση ε, από εσά. Τι μπορούμε να πούμε στους πολίτες αυτούς που μου ζήτησαν τη γνώμη μας. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε ε, και αν ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο σε αυτό τον τομέα. Εάν ε, αποκτήσω ένα οικόπεδο ή ένα σπίτι, ε, εφόσον έχω πληρώσει για αυτό το οποίο ε, αποκτώ, δεν μπορεί να έρθει το κράτος και να πει ότι δεν είναι δικό μου και πρέπει να πληρώσω κάποιους φόρους επιπλέον. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στους πολίτες και γι' αυτό θα ήθελα να σα ζητήσω τη στήριξή σα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε του πολίτε. Thank Κύριε ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για την έκθεση αυτή. Εκτιμώ ιδιαίτερο την προσέγγισή σας. Παίρνετε συγκεκριμένα παραδείγματα προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινή ζωή τους και προσπαθείτε να άρετε τους φραγμούς ε, και χαιρετίζουμε την προσέγγιση αυτή. Μερικές φορές όμως δεν αρκεί το να άρουμε τους φραγμούς για να δώσουμε στους πολίτες της Ευρώπης και την αίσθηση του ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω αυτά τα θέματα ηθαγένειας που είναι γνωστά σε όλους και που νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσετε στο πλαίσιο της συζήτησης για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ένα θέμα είναι η αγορά εργασίας. Δεν μπορεί κανείς να μετακινηθεί ελεύθερα στην Ευρώπη με την οικογένειά του ή να αγοράσει αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο αν δεν έχει το δικαίωμα να εργαστεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και γνωρίζετε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν περιορισμοί χωρίς να, υπάρχουν, να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι η μόνη που μπορεί να πιέσει τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον να δίνουν κάποια αιτιολόγηση. Ένα δεύτερο θέμα που αφορά και τον ε, τρόπο με τον οποίο μας βλέπουν οι άλλοι εμάς τους Ευρωπαίους. Γιατί αν ε, μας κοιτάξει κανείς με τη ματιά ενός Αμερικανού υπαλλήλου που πρέπει να δώσει θεώρηση διαβατηρίου σε ένα Ευρωπαίο πολίτη που θέλει να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, σαφώς υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν λέω ότι είναι δικό σα θέμα, δική σα αρμοδιότητα, Πάντω, σαφώ εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να το διαπραγματευτεί εκ μέρου όλων μα με τρίτε χώρε για τέτοια θέματα, όπω το καθεστώ θεώρηση διαβατηρίου. Αυτά τα δύο σημεία λοιπόν ήθελα να, να σας αναφέρω και να τα λάβετε υπόψη σα, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιαίτερα τολμηροί και παλεύετε και δίνετε μάχες εκεί που άλλοι τα παρατάνε. Ευχαριστώ, κύριος Μαρτίνεφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο και την Πρόεδρο της Επιτροπής. Θέλω καταρχήν να σας συγχαρώ για την έκθεσή σας και για την παρουσίαση που μας κάνατε σήμερα. Θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι έχετε την υποστήριξη όλων μας για πολλές προτάσεις που συμπίπτουν με τις δικές μας ανησυχίες και ανάγκες. Δεν θέλω να επαναλάβω θέματα που ήδη συζητήθηκαν. Αλλά θέλω να αναφερθώ σε ένα σημείο που εσείς δεν αναφέρατε. Το θεωρώ όμως κέρια σημασίας όταν θέλουμε να δείξουμε στους πολίτες ότι υφίστανται τα δικαιώματά τους. Τα έγγραφα που μας μοιράσατε τα είδα και μου φαίνονται χρήσιμα και σημαντικά. Θα ήθελα όμως να μιλήσω ως Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου υπεύθυνο για την πολυγλωσία. Νομίζω ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι πραγματικά χρήσιμο. Μπορεί να μας καθησυχάζει, αλλά δεν το εκδίδουμε σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμο, γιατί οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλούν όλες τις γλώσσες και εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και θα ήθελα να ακούσω τις προθέσεις σας επ' αυτού. Πιστεύουμε, όπως πιστεύει η Επιτροπή για την καθημερινή της δουλειά, ότι με τρεις γλώσσες καλύπτονται οι ανάγκες μας. Δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε όμως το ευρύ φάσμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους θέλουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε για τα δικαιώματά τους και δεν βλέπω να έχει γίνει πρόοδος επ' αυτού. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις προθέσεις σας και να ακούσω τι δεσμεύσεις αναλαμβάνεται ούτως ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για τη δουλειά που γίνεται για τα δικαιώματά τους. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε τους πολίτες, στους πολίτες στη γλώσσα τους, όχι μόνο σε δύο ή τρεις γλώσσες. Θα στοχίσουμε, δεν θα επιτύχουμε κατά κανένα τρόπο το στόχο μας εάν περιοριστούμε στις δύο ή τρεις γλώσσες. Πείτε μου λοιπόν Ποιες είναι οι προθέσεις σας για αυτό το θέμα. Αφορά τη δημοσίευση εγγράφων και, και ανακοινώσεων της Επιτροπής που πρέπει να φτάνουν σε όλους τους πολίτες, σε όλες τις γλώσσες. Διαφορετικά, εάν δεν μπορέσει να το διαβάσει και ο Σλοβαίνος και ο Σλοβάκος και ο Ισπανός και οποιοδήποτε πολίτη στη γλώσσα του, δεν φτάνουμε κοντά στον πολίτη. Ξέρω ότι δεν είναι φτηνό είναι ίσως πολύ πιο δαπανηρό από ό,τι κάποιοι πιστεύουν. Χθε στην Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε το σχόλιο μιας Γερμανή συναδέλφου που είπε ότι θα πρέπει να εργαζόμαστε μόνο σε δύο-τρεις γλώσσες. Διότι όντως είναι ε, ακριβό αυτό που κάνουμε. Και τη ρώτησα, ξέρετε πόσο κοστίζει η γλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντω κανένας από όλους τους συναδέλφους ήταν παρόντες, από όλους τους παριστάμενους συναδέλφου, κανένα δεν ήξερε. Κανένα δεν ήξερε ότι η πολυγλωσία σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοστίζουν λιγότερο από την τιμή ενός καφέ για κάθε πολίτη της Ένωσης το χρόνο. Πολύ φθηνά λοιπόν. Και πολύ λίγα πράγματα κοστίζουν λιγότερο από ένα καφέ αναπολίτη μία φορά το χρόνο. Ξεκινώ βεβαίως από την ε, ε υπόθεση ότι αν είμαστε 500 εκατομμύρια ε, πολίτες κοστίζει η πολυγλωσία 500 ε, εκατομμύρια ευρώ. Όταν λοιπόν λέγεται ότι πρέπει να δουλεύουμε σε δύο γλώσσες, καλά θα είναι εάν ε, ο καθένας μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα του. Εάν ε, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι μπορούν να μιλούν τη γλώσσα μου όπως εγώ μιλάω γαλλικά και γερμανικά, έχει καλό. Ας το κάνουμε τότε έτσι όλοι, για να είμαστε όλοι στην, ε, σε, στην ίδια κλίματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνετε λοιπόν μια προσπάθεια ώστε ό,τι κάνετε ως ανακοίνωση κάνουμε εδώ, να μπορεί να δημοσιεύεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε όντως να μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο, πρόοδο την οποία αξίζει η δουλειά που, που επιτελείται. Διαφορετικά, πραγματικά όλα αυτά θα περιορίζονται σε κάποιους πολύ περιορισμένους κύκλους και δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την πρόοδο που θέλουμε. Και πάλι τελειώντας θα σας ευχαριστώ την εκκλησία σας κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Γιάρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την έκθεση και τις επεξηγήσεις σας κυρία Επίτροπε. Εξαιρετική ιδέα το 2013 να γίνει το έτος των πολιτών, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτός σκοπός, υφίσταται για τους πολίτες της. Και στην πολιτική θέτουμε προϋποθέσεις πλαίσιο μόνο και είναι καλό να κινούνται εκεί οι πολίτες. Υπάρχει συνεχώς ένας διάλογος μέσα σε αυτά τα πλαίσια Άλλωστε και στην Επιτροπή Αναφορών βλέπουμε ότι οι πολίτες προσφεύγουν σε μας όταν είναι δυσαρέστημένοι και όταν έχουν διαφορετικές προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει από την άλλη ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Αναφερθήκατε σε ορισμένα βασικά θέματα, συμφωνώ. Πιστεύω βέβαια ότι πρέπει να προσπαθήσουμε κι άλλο βασικός κανόνας. Πρέπει οι ρυθμίσεις να εφαρμόζονται, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες, αλλά και οι διοικήσει στα κράτη-μέλη πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες. Στην Επιτροπή Αναφορών βέβαια με ενδιαφέρει τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να λειτουργήσουν ταχύτερα οι διαδικασίες. Πολλές φορές έχουμε ε, διαπιστώσει προβλήματα Πολλές φορές δεν τηρούνται οι κανόνες, διαπιστώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά περνάει πολλής χρόνος μέχρι ότου πάρει μπρο η διοίκηση του κράτους μέλους και όντως σεβαστεί το, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει να επιταχύνονται. Επίσης, πού πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες. Μιλήσατε για ελεύθερη κυκλοφορία, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο και περισσότερο αυτονοήτως αξιοποιούν το δικαίωμα αυτό με ταξίδια, μεταξύ άλλων, αλλά όλο και περισσότερο πηγαίνουν να εργαστούν αλλού, όχι μόνο να ταξιδέψουν, εγκαθίστανται αλλού. Θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, εκλέγην και εκλέγεστε. Αυτό είναι πολύ θετικό. Δηλαδή δεν θέλει μόνο να δουλέψει αλλά και να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι συμμετέχει στη διαμόρφωση της περιφερειάς του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του αυτό. Επίσης, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Αγορά. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι ήδη. Εκεί ο πολίτης έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο από την υφιστάμενη πολιτική ως προς τις προσδοκίες του. Δηλαδή περιμένει ότι η ιδιοκτησία θα είναι σεβαστή παντού και θα υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την απόκτηση ιδιοκτησίας αλλά και τις αποζημιώσεις σε περίπτωση απαλωτρίωσης για παράδειγμα. Πολλές φορές ε, εδώ φτάνουμε στα όρια μας, γιατί υπάρχει το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά μας λένε ότι υπάρχει και το, το εσωτερικό δίκαιο του κράτους μέλους. Και τι να κάνουμε. Ο πολίτης όμως ε, τα βλέπει τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μπορεί να λέμε ότι συνδέονται αυτά, ούτε ο πολίτης ε, θα ικανοποιηθεί αν δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από μια καθαρά νομική απάντηση. Επίσης, κάτι ακόμα. Η Επιτροπή Αναφορών ασχολήθηκε πολύ με κάτι άλλο. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα θέλουν οι νομικές πράξεις ενός κράτους μέλους να αναγνωρίζονται από ένα άλλο κράτος μέλος. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Να, συζητήσαμε σήμερα για τους ε, γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Άλλες φορές είχαμε προβλήματα με το δίκαιο υιοθεσίας ε, διότι μια απόφαση σε ένα κράτο μέλος δεν αναγνωριζόταν από ένα άλλος, άλλο. Συγγνώμη. Οπότε, για να τελειώνω, θεωρώ το έργο σας ιδιαίτερα σημαντικό και είναι πάρα πολύ καλό ο πολίτης και είναι μια γόνιμη διαδικασία αυτή να συμβάλλει και ο πολίτης στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ε, δικαίου, γιατί πολλές φορές ο πολίτης σκέφτεται πιο προχωρημένα από τους πολιτικούς. Ευχαριστώ, Μποτσινάρο Άουκεν. Σύντομα, παρακαλώ, για να μπορεί και να έχει την ευκαιρία η Επίτροπος να απαντήσει. Ευχαριστώ. Επίτροπε και την Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Όπως συνήθως, μου κάνει εντύπωση και το περιεχόμενο και η ποιότητα της παρουσίασής σας. Αλλά επειδή πάντα ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας πω, Επιτρόπε, ότι ένας Γάλλος γιατρός, υπήκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το επάγγελμά του ή ένας καθηγητής πανεπιστημίου. δεν έχει ένας καθηγητής πανεπιστημίου από τη Βρετανία, παραδείγματο χάρη, δεν έχει τα ίδια δικαιώματα όπως ένα συναδελφός του στην Ιταλία. Είναι παραδείγματα που, τα έχουμε δει στην πράξη, διακριτική μεταχείριση κατά πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί τη βάση της εθνικής τους καταγωγής. Και πρόσφατα είπατε και εσείς οι ίδια, κυρία Επίτροπε, ότι φτάνει πια είπατε enough is enough. Και μετά ε, υπάρχει το θέμα της αναγνώρισης των δικαιωμάτων. Κάτι που δεν είναι δεδομένο για όλους τους πολίτες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διαδικασίες παραβίασης του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων, κάτι το οποίο δημιουργεί εμπόδια σε πολλούς από τους πολίτες μας. Τέλος, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από λίγες εβδομάδες κάναμε μια έντονη και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Στρασβούργο σχετικά με την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, ε, κάτι που έχει σχέση με τις Ευρωπαϊκές Ένωσης ε, ε, και καθώς ε, μας έδωσε την ευκαιρία η Ουγγρική Προεδρία να συζητήσουμε πάρα πολύ το θέμα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε, αν συμφωνείτε με την επίσημη θέση της Επιτροπής, που ζήτησε από την Ουγγαρία να επανεξετάσει την ομοθεσία της για θέματα μέσων ενημέρωσης και αν θα κάνετε την ίδια κίνηση και προς τη Ρουμανία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη Ρουμανία. Θα ήθελα να σας πω ότι στη Ρουμανία οι μυστικές υπηρεσίες δηλώνουν την παρουσία τους και ανησυχούν και τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς στην Ρουμανία σχετικά με την ελευθερία του τύπου και μπορώ να σας δείξω συγκεκριμένα έγγραφα που δείχνουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ρουμανίας ε, επισκέφθηκαν τη δική μου ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Έχουν ε, υπάρξει πάνω από 100 επισκέψεις στην ιστοσελίδα μου και επιβεβαιώθηκε ότι η διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε είναι η, διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση των, των μυστικών υπηρεσιών. Εάν αυτό συμβαίνει στην ιστοσελίδα ενό βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φανταστείτε τι γίνεται για του δημοσιογράφου. Κυρία Άουκεν, θα μιλήσω αγγλικά και όχι δανέζικα. Και έχει σχέση αυτό που θέλω να πω με αυτό που είπε και ο κύριος Ποστινάρου. Και είμαι βεβαίω ότι μπορείτε να απαντήσετε γιατί έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ στην Επιτροπή μας σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, σχετικά με το αν το όλο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να ισχύσει για το ευρωπαϊκό δίκαιο ή όχι. Το ερώτημα της ελευθερίας του τύπου και των μέσων ενημέρωσης και στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία και η διακριτική μεταχείριση είναι ένα θέμα για το οποίο αναγράφεται στη συνθήκη ότι ο χάρτης δεν διευρύνει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα κρατών μελών. Όμως, επίσης αναγράφεται σαφώς το άρθρο 7 ότι η διακριτική μεταχείριση και η ελευθερία του τύπου ε, είναι δικαιώματα που όταν παραβιάζονται Υπάρχουν διάφορες κλιμακούμενες δυνατότητες που αναγράφονται στο άρθρο 7. Μετά τη συζήτηση που κάναμε και σήμερα, εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκινήσαμε πριν από μήνες ή και χρόνια όταν ακούσαμε ότι δεν ισχύουν τα κριτήρια της Κοπενχάγης από τη στιγμή που είναι ένα κράτος, κράτος μέλος αλλά δεν είναι αποδεκτό αυτό για τόσο θεμελιώδη δικαιώματα όπως είναι η ελευθερία του τύπου. Σε συγκεκριμένες χώρες υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι ε, για τους, με τους οποίους πρέπει να ασχοληθεί το δικαστήριο στο Στρασβούργο, αλλά χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε τις βασικές αξίες του άρθρου 2 και να μην παραβιάζονται τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 7, το οποίο τώρα είναι πιο χρήσιμο από ό,τι στο παρελθόν. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί μπορεί και το Κοινοβούλιο αλλά και η Επιτροπή των Τρίτων των Κρατών Μελών να επισημάνουν ότι κάτι πάει στραβά και μετά θα χρειαστούν τα 4 πέμπτα των κρατών μέλων για κάτι σοβαρότερο. Αλλά όπως και εσείς το κάνατε στην περίπτωση της διακριτικής μεταχείρισης κατά τον Ρωμά, και εγώ είμαι ε, απολύτως υπέρ αυτών που είπατε. Άκουσα πολύ προσεκτικά τι είπατε. Είπατε ξεκάθαρα, δεν είπατε ότι είναι σαν αυτό που έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είπατε ξεκάθαρα, φανταστείτε να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μετά από αυτά που συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και άκουσα ότι στρεβλώθηκαν αυτά που είπατε, που παρομοιάστηκαν ε, τα λόγια σας, σαν να είχατε πει ότι αυτά που έγιναν, παρόμοια με αυτά που έγιναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά όμως δεν ήταν πολύ ξεκάθαρα ε, ε, αυτά τα οποία ε, ακολούθησαν και ακριβώς είναι η θέση. Και ήταν πιο ευέλικτη η ερμηνεία που ακούσαμε αργότερα από τις, στις προηγούμενες απαντήσεις που είχαμε πάρει από την Επιτροπή είναι θέματα που αφορούν ε, τα μέσα ενημέρωση τα δικαιώματα ιδιοκτησία, τη διακριτική μεταχείριση και είμαι πολύ περίεργη αν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά ή όχι, γιατί θα ήταν κρίμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορούμε να ασχοληθούμε εμεί με τέτοια θέματα. κυρία Μπασέσκου, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θέλω να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Μποστινάρου για την αναφορά για την ελευθερία τύπου στη Ρουμανία. Διευκρινίζω ότι στη Ρουμανία δεν υπάρχει νόμος που να ρυθμίζει την ελευθεροτυπία. Υπάρχει μια στρατηγική ασφαλείας που έχει ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται σε κατά παραγγελία αν θέλετε ε, εκστρατείες στον τύπο. Διότι αυτές ε, κατά ανάθεση οι εκστρατείε στον τύπο υπάρχουν από διάφορες εταιρείες ή οργανισμούς για να ασκήσουν πίεση. Η περίπτωση της Ρουμανίας δεν έχει σχέση με την περίπτωση της Ουγγαρίας. Το λέω αυτό σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Μπουστινάρο. Ευχαριστώ. Και τώρα η Επίτροπος, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είπαμε από την αρχή ότι υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός που μας έκανε να καθυστερήσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν γραπτός από εμένα γιατί δεν θα προλάβουμε. Υπάρχουν όμως δύο ερωτήσεις που θέλω να τις καταπιαστώ τώρα γιατί Πολλές σκέψεις έχουν γίνει σε σχέση με το που βρισκόμαστε και προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Οπότε χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις από την πλευρά μου. Στην ερώτηση για τις γλώσσες πρώτα απ' όλα, γιατί η δυσαρεστημένη εδώ είμαι εγώ, η μόνη που δεν μπορώ να μιλήσω τη λουξεμβουργική μου μητρική γλώσσα. Την παρισμένη εβδομάδα ήταν η 20η επέτειος μιας πολύ σημαντικής αναφοράς σχετικά με τη χρήση των καταλανικών. Και εγώ ήμουνα η συντάκτρια, γι' αυτό θυμάμαι και αναφέρθηκε από τον καταλανικό τύπο 20η επέτειος, που ήταν πολύ σημαντική αναφορά, γιατί έθεσε επιτάπητο στο θέμα της προσέγγισης μας των διαφόρων γλώσσων, στις διάφορες γλώσσες. Πώς αντιμετωπίζουμε τις γλώσσες. Τότε είχαμε να κάνουμε με μία μη επίσημη γλώσσα. και όμως ως Λουξεμβούργια λέω ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μεγάλων και μικρών γλωσσών. Υπάρχουν μητρικές γλώσσες μόνο και η μητρική γλώσσα του καθενός είναι η ωραιότερη του κόσμου. Κατόπιν τούτου βέβαια πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και να χρησιμοποιούμε γλώσσες εδώ στους, στα διεθνή όργανα και στους διεθνείς οργανισμούς που μας επιτρέπουν να εργαζόμεθα. Και πάω στους πολίτες τώρα. Οι γλώσσες που μιλούνται στην περιφέρεια όπου ζουν οι πολίτες, οι γλώσσες στις οποίες εκφράζονται οι πολίτες. Αυτά σκεφτόμαστε όταν πριν από 20 χρόνια αποφασίσαμε υπέρ της χρήσης των καταναλικών στην Καταλωνία, στα γραφεία ε, ενημέρωσης και τύπου μας. Δηλαδή, με ρεαλιστικό τρόπο, όχι με ιδεολογήματα, αλλά αναφερόμενοι στα προβλήματα των πολιτών και μιλώντας τους στον τόπο τους, στη γλώσσα τους. Ε, σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι προχωρούμε σε αναδιοργάνωση των γραφείων μας στις χώρες μέλη και υπάρχουν σαφείς οδηγίες να χρησιμοποιούν τη γλώσσα του τόπου και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα και που γίνεται κατανοητή από τους πολίτες. Οπότε δεν αλλάξαμε την προσέγγιση μας και με μένα ως επίτροπο στο θέμα αυτό να είστε σίγουροι ότι πάντα η πολυγλωσία είναι σημαντική στην ημερησία διάταξη. Τώρα, τι άλλε ερωτήσει ερωτήσεις δεν θα τις απαντήσω, προσπερνώ πολλέ δηλαδή, για να απαντήσω γραπτό. Πάω τώρα στην εφαρμογή του χάρτη, γιατί αυτό έχει σχέση με πολλές από τις ερωτήσει σα. και πράγματι υπάρχει μια σάφια. Τον Οκτώβριο, πέρσι, παρουσίασα μία ανακοίνωση για την ε, αντικειμενική εφαρμογή του χάρτη στον τρόπο εργασίας μας. Και στην ανακοίνωση εκείνη έκανα, προέβλεψα έναν έλεγχο όλων των νομοθετημάτων που προτείνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο οικονομική ανάλυση των επιπτώσεων μιας νομοθετικής πρότασης, αλλά και μια ανάλυση των επιπτώσεων που η πρόταση αυτή θα έχει στις αρχές που ε, υπάρχουν στο χάρτη. Και μπαίνω στον πυρήνα του θέματος. Ο χάρτης είναι σαφές. Εφαρμόζεται μόνο όταν θεσπίζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία και όταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία, το ευρωπαϊκό δίκαιο εφαρμόζεται στα εθνικά κράτη. Δηλαδή δεν υπάρχει οριζόντια εφαρμογή. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό, όχι ε, από τους βουλευτές εδώ, αλλά από τον απλό κόσμο που λέει υπάρχει χάρτης και κοιτάξτε εδώ που δεν τον εφαρμόζουν το χάρτη. Γιατί κανείς δεν εξήγησε ότι οι κυβερνήσεις δεν ήθελαν την οριζόντια εφαρμογή του χάρτη. Γιατί αν το ήθελαν κάτι τέτοιο δεν θα συμπεριελάμβαναν το άρθρο 51 στους κανόνες μας. Ορίστε λοιπόν, μπορούμε να εφαρμόζουμε το χάρτη όταν νομοθετούμε ή ελέγχουμε ή εφαρμόζουμε την ομοθεσία. Ας πάρουμε το Ρωμά. Το πρόβλημα των Ρώμα συνδέθηκε προς την οδηγία του 2004 για την ελεύθερη κυκλοφορία και την μη εφαρμογή στη γαλλική νομοθεσία για των ε, δικονομικών δικαιωμάτων ενός προσώπου για να προστατευτεί το άτομο αυτό ε, απέναντι στην ε, αυθαίρετη συμπεριφορά ενός κράτους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Σε αυτό το επίπεδο είμαι υπεύθυνη εγώ για την ελεύθερη κυκλοφορία και σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσα να ζητήσω από την Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Γαλλίας, την οποία αναστήλαμε τη διαδικασία γιατί η Γαλλία υποσχέθηκε ότι την άνοιξη τούτου του έτους θα προχωρήσει σε μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της. Ουγγαρία. Ο νόμος για τα ΜΜΕ. Το ίδιο πάλι. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός νόμος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ως Επίτροπος έπρεπε να το εξηγήσω αυτό το 2009 στο Ινολομέλεια. Και θυμάστε τι έντονη συζήτηση ήταν εκείνη και βέβαια τότε δεν σας ευχαρίστησα βέβαια, τότε δεν υπήρχε ο χάρτης. Αλλά ήδη ήταν σαφές ότι δεν είχαμε, δεν έχουμε και μάλλον και δεν θα έχουμε ευρωπαϊκό νόμο για τα μιμία. Έχουμε την οδηγία για τις ε, οπτικοακουστικές υπηρεσίες χωρίς σύνορα, που, ήταν, που είναι η διάδοχος της τηλεόρασης χωρίς σύνορα. Οπότε, μόνο εδώ έχουμε, όχι για τα μημία. Η Επίτροπος υπεύθυνη για τα οπτικοακουστικά ήταν και εκείνη που παρενέβη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτό είναι το μόνο συγκεκριμένο που έχουμε στα χέρια μας. Μόνο με βάση αυτό μπορούμε να ε, κατηγορήσουμε μια κυβέρνηση για την ελληπή εφαρμογή της οδηγίας. Και για όσους σε όσους δεν θυμούνται, θα θυμίσω ένα γεγονός. Είχα προτείνει ως επίτροπος τηλεπικοινωνιών και οπτικοακουστικών τότε να προσθεθεί άρθρο στη νέα οδηγία σχετικά με την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων στα ΜΜΕ. Αυτή ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 24 κράτη-μέλη καταψήφισαν την πρόταση. Η Βρετανία, η Ολλανδία και η Λετωνία δεν καταψήφισαν, έτσι για να ξέρετε ποιοι καταψήφισαν. Και μετά τις πιέσεις του Κοινοβουλίου προσθέθηκε μια θεολογική σκέψη, αν θυμάμαι καλά, που τι να κάνει, δεν έχει νομική ισχύ μεγάλη θεολογική σκέψη, αλλά σας τα λέω. Ήταν σαφές ότι σε εκείνο το επίπεδο η Επίτροπος υπεύθυνη για τα ΜΜΕ, τα οπτικοακουστικά, ε, έπρεπε να παρέμβει και να απευθύνει επιστολή στις αρμόδιες αρχές για να ζητήσει από τις αρχές να αλλάξουν στο εσωτερικό δίκαιο αυτά τα ε, στοιχεία που δεν συμφωνούσαν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Σας τα λέω αυτά για να εξηγήσω πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Και περνάμε έτσι στο μεγάλο πρόβλημα που εντοπίσατε πολλοί από εσάς ότι δεν γίνονται κατανοητά όλα αυτά από τρίτους, από ανθρώπους που δεν είναι στα θεσμικά όργανα. Το άρθρο 7 είναι πυρηνική βόμβα. Ε, εντάξει, να, να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά πραγματικά είναι μια ατομική βόμβα που χρησιμοποιείται αν υπάρξουν τεράστια προβλήματα σε κάποιο κράτος μέλος. Η Νέλη Κρούζ, επίτροπος υπεύθυνη για τα οπτικοακουστικά, είπε ότι θα εξετάσει το θέμα και πάω έτσι στο ζήτημα της Ρουμανίας. Είπε λοιπόν ότι θα εξετάσει την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη σε σχέση με την μη εφαρμογή, την ελλειπή εφαρμογή των, ε, της οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Οπότε θα τα δει αυτά με τρόπο οριζόντιο. Αυτό δεν είναι το πρόβλημά μας εν προκειμένου βέβαια. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το χάρτη ο οποίος οριζόντια εφαρμογή δεν μπορεί να έχει. Και Περνάω έτσι και στο ισπανικό ερώτημα σχετικά με το δίκαιο ιδιοκτησίας που εμπίπτει σε αυτό το πρόβλημα. Έχω ήδη απευθύνει τη δεύτερη επιστολή μου προς τους Ισπανούς ομολόγους μου για αυτό το ζήτημα. Αν δεν μπορούμε να αποδείξουμε τη σαφή διακριτική μεταχείριση Ευρωπαίων πολιτών σε σύγκριση με τους Ισπανούς πολίτες. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά οι πολίτες ενίστανται και λένε ναι αλλά εμείς έχουμε δικαιώματα βάσει του χάρτη. Και τι θα τους απαντήσουμε, μάλιστα. Θα τους απαντήσουμε ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι πολίτες ε, της χώρας και προσφεύγουν, μπορούν να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια και αφού προσφύγουν και εξαντλήσουν όλες τις ε, δυνατότητες, τότε θα απευθυνθούν στο Στρασβούργο, στο ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για αυτά. Δεν μπορούν όμως να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, αφού ο χάρτης δεν ε, εφαρμόζεται. Δηλαδή δεν ισχύει αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία ή ευρωπαϊκός κανονισμός που να προβλέπει την εφαρμογή του. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα το λύσουμε, γιατί χρειάζεται η τροποποίηση της συνθήκης. Γιατί τώρα ξέρετε ότι είμαστε στην διαδικασία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει μέλος ή θα προσχωρήσει στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και μπορώ να σας πω ότι οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται θετικότατα και την Άνοιξη θα ολοκληρωθούν, όπως ελπίζουμε με τρόπο πολύ θετικό. Θα βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των δύο δικαστηρίων, οπότε εξελίσσονται καλά τα πράγματα. Μετά θα περάσουμε μια μακρά διαδικασία κυρώσεων, ε, επικυρώσεων, αλλά αυτό δεν λύνει το ε, πρόβλημα, το οποίο παραμένει ακριβώς το ίδιο. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτό το κανάλι πάλι δεν βρίσκεται λύση. Το λέω αυτό για όλους όσου λένε εντάξει, αλλά όταν θα ε, με την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν θα λυθεί. Αν αποφασίσει το δικαστήριο του Στρασβούργου, θα βρεθεί ότι οι οδηγίες μας δεν συμφωνούν με τις αρχές για των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει και το προηγούμενο σε σχέση με το άσυλο και τη μετανάστευση. Άρα χρειάζεται τροποποίηση της συνθήκης και θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 51 του χάρτη αν θέλουμε να υπάρξει αυτή η σαφήνεια που την θέλουν όλοι και η οποία όμως σαφήνεια σε δεν έχει νομική ισχύ, δεν υφίσταται νομικά. Διαβάστε την ανακοίνωση του Οκτωβρίου που το διευκρινίζει αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάθε φορά που υποβάλλουμε νομοθετικές προτάσεις λαμβάνουμε υπόψη μας το χάρτη και κάθε φορά ελέγχουμε αν η ευρωπαϊκή νομοθεσία εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Πάντα έχουμε υπόψη μας και τον χάρτη, αλλά κατά τα άλλα ισχύει η επικουρικότητα. Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε, αλλά αυτά είναι τα νομικά ε, γεγονότα. Τώρα, για τα υπόλοιπα και για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέσατε, επειδή δεν προλαβαίνω να απαντήσω, θα λάβετε απάντηση γραπτός. Όμως το πλαίσιο που παρουσίασα τώρα παραμένει ίδιο και ισχύει για όλες τις ερωτήσεις που υποβάλατε. Τις αφορά όλες τις ερωτήσεις σας. Επίσης, παλιά δύσκολα πίστευαν ότι ο χάρτης θα γίνει πραγματικότητα και πολλοί που διαπραγματεύτηκαν το χάρτη ξέχασαν τι διαπραγματεύτηκαν. Αυτό ισχύει και για τα κράτη-μέλη. Αλλά και εδώ στο Κοινοβούλιο, επειδή δεν υπάρχουν πια ακόμη οι βουλευτές που συμμετείχαν στην ε, ε, συνέλευση και που θυμούνται τις, ε, το σκεπτικό και τις εξελίξεις που είχαμε ακολουθήσει τότε γιατί φτάσαμε στο άρθρο 51, δεν θυμούνται. Ας αξιοποιήσουμε το καλύτερο που, από τους κανόνες που έχουμε. Έχει βελτιώσει ο χάρτης πάρα πολύ την κατάσταση σε σχέση με την προτέρα, προχάρτη δηλαδή. Ας τον εφαρμόσουμε λοιπόν με τρόπο θετικό. Μιλάμε για δίκαιο, για τον, τους νόμους. Αυτό που θέλουν να ξέρουν οι πολίτες είναι τι κάνουμε συγκεκριμένα για την επίλυση των προβλημάτων τους. Δεν τους νοιάζουν όλα αυτά τα, αυτοί νομικοί συλλογισμοί. Έχω συμμετάσχει σε πολλές προεκλογικές εκστρατείες και ξέρω πώς ε, σκέπτονται και αντιδρούν οι πολίτες. Χαίρομαι λοιπόν που άκουσα από όλους σας και από όλα τα κόμματα, γιατί έχω πάει και σε άλλες επιτροπές όπου η αντίδραση δεν ήταν όπως η δική σας. Εγώ χαίρομαι γιατί όλοι αναγνωρίζετε την ανάγκη για το έτος των πολιτών, όχι για την ηθαγένεια, γιατί η ηθαγένεια έχει να κάνει με τα εθνικά κράτη και τις αποφάσεις τις εθνικές. Το έτος των πολιτών λοιπόν, γιατί εσείς τους αντιμετωπίζετε άμεσα τους πολίτες. Βοηθήστε με λοιπόν να κάνω το έτος αυτό ένα χρήσιμο εργαλείο που θα μπορώ να χρησιμοποιώ και όλοι μας για να εξηγούμε στους πολίτες μέχρι που φτάνουν τα δικαιώματά τους. Συμφωνώ με την ανάλυση σας ότι αν στραβώσουν τα πράγματα και αν Ε, δεν συγκεντρωθούν οι πλειοψηφίες, ε, δεν διαμορφωθούν οι συσχετισμοί που πρέπει, πάντα υπάρχει αυτή η ατομική βόμβα το άρθρο 51. Καλά, ε, μην πάμε αμέσως στην ατομική βόμβα, υπάρχουν και τα καλά σνικοφ. Όχι, αλλά εννοώ ότι κανείς Δηλαδή υπάρχει απειλή, υπάρχουν οι, οι Την απειλή έψαχνα. Η απειλή δηλαδή των κυρώσεων της ατομικής βόμβας, εάν κάτι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει και αυτό. Έτσι. Να φυλάγεστε λοιπόν από τα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Και έχετε δίκιο στην ανάλυση σας για τα κριτήρια της Κοπενχάγης, έτσι όπως ε, προχωρούμε βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν και κάποια παράλογα στοιχεία. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα αλλάξουμε, τα εξαλείψουμε και να αξιοποιήσουμε τους κανόνες μας με το βέλτιστο τρόπο. Να πω κάτι άλλο για να μην τελειώσω με αρνητικά σχόλια και σκέψεις. Εγώ είμαι η επίτροπος εκείνη που είναι η πλέον ευτυχής με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας ήταν αδιανόητον να δημιουργηθεί η Ευρώπη της δικαιοσύνης, μια ήπειρος δικαιοσύνης. Από κοινού προχωρήσαμε σε αυτό το θέμα ανέλπιστα γρήγορα και καταφέραμε βήμα το βήμα σταδιακά να βάλουμε όλα τα στοιχεία επιτάπητος και να αποφασίσουμε σε χρόνο ρεκόρ. Και πρέπει να το πούμε στους πολίτες ότι προχωρούμε σε ό,τι αφορά το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε για το 2012 και να βγούμε στους πολίτες το 2013 και να τους εξηγήσουμε πολύ συγκεκριμένα τι κάνει η Ευρώπη για αυτούς. Μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά μπορούμε μέχρι τότε να κάνουμε πολλά. Πρέπει να τα εξηγήσουμε όλα στους πολίτες και να τους δώσουμε την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ένωση για την οποία μπορεί να είναι ε, περήφανοι. Θα μιλήσω γαλλικά για να μιλήσω και μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας σας. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω τα έγγραφα αυτά να τα δημοσιεύσετε και στα καταλανικά για να τα διανύμουμε στην Καταλωνία. Αλλά δεν θα αγνοείτε ότι οι δύο επίσημες γλώσσες στην Καταλωνία είναι οι επίσημη γλώσσα στην Καταλωνία είναι δύο. Κανένας Καταλανός δεν αγνοεί τα Ισπανικά. Αντιθέτως υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια που ζουν στην Καταλωνία και δεν ξέρουν Καταλωνικά. Πρέπει να σας πω ότι άτομα της δικής σας πολιτικής ε, οικογένειας ήταν αντίθετοι στο να γίνει επίσημη γλώσσα η καταλανική. Σας ευχαριστώ και να σας πω αυτά που έχω να πω για να καταλάβει κανείς και να ακούσει τους πολίτες, πρέπει να τους καταλάβει και να το ακούσει τη γλώσσα του. Colleghi, scusatemi, io vorrei riprendere i lavori prima. Αγαπητοί συνάδελφοι, Dobbiamo esaminare la petizione. Περνούμε τώρα στην αναφορά αριθμός 1746 του κύριου Μαξίμ Ρεβά. Δεν είναι παρόν αναφέρον. Θα δώσω το λόγο στην υπεύθυνη της Επιτροπής, την εκπρόσωπο τη Επιτροπή ή στον υπεύθυνο, στον κύριο Τύπο Μπαζή. Έχουμε την αναφορά του κυρίου Μαξίμ που αφορά το δικαίωμα του εκλέγην ατόμων που ζουν στην Εστονία και δεν έχουν απροσδιόριστη ηθαγένεια. Μιλούμε για δικαίωμα του εκλέγην σε εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναφέρθηκε στην αναφορά του ότι τα άτομα αυτά που ζουν στην Εστονία και έχουν τη ηθαγένεια δεν έχουν το δικαίωμα εκλέγην στις ε, εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πράγμα το οποίο, κατά τον αναφέροντα, οδηγεί σε δημοκρατικό έλλειμμα και λέγει ότι η αρχή της μη πρέπει να θεωρείται γενική αρχή της κοινωτικής νομοθεσία. Αυτό ζητεί λοιπόν ο αναφέρον να επιτραπεί σε αυτά τα άτομα να συμμετέχουν σε εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας πω σύντομα ποια ήταν η απάντηση της Επιτροπής γραπτός. Όντως, η Επιτροπή γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Απ' την άλλη όμως, δεν πρόκειται για ένα νέο θέμα, δεδομένου ότι και το θέμα και στο παρελθόν και εκφράστηκαν κάποιες ε, ανησυχίες. Αυτό αποτέλεσε και αντικείμενο κάποιων ερωτήσεων που απέφθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις απαντήσεις της πάντα η Επιτροπή έλεγε ότι έχουν ε, καταβληθεί στο παρελθόν προσπάθειες και κυρίως κατά τη διάρκεια στην προενταξιακή στρατηγική ώστε να μπορέσουν τέτοιου είδους άτομα να πάρουν την ηθαγένεια της χώρας στην οποία διαμένουν αλλά θα πρέπει από την άλλη πλευρά να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι συνθήκες για την ε, χορήγηση της ε, ηθαγένειας ή για την απόλυτη της ηθαγένειας από κάποιον είναι θέμα της απόλυτης δικαιοδοσίας κάθε κράτους μέλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερη να ορίσει τους όρους τους οποίους κάποιος παίρνει την ηθαγένεια Σύμφωνα με την γενοτική νομοθεσία λοιπόν δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από νομικής πλευράς τέτοιου θέμα. Τώρα, όσον αφορά το δικαίωμα του εκλέγην, και εδώ είναι περιορισμένες οι αρμοδιότητές μας, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Το κοινοτικό ε, δίκαιο χορηγεί δικαιώματα του εκλέγην στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ευρωπαϊκές εκλογές και μπορούν να ψηφίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ή στην χώρα καταγωγή ή στη χώρα διαμονής τους. Αυτά όμως τα εκλογικά δικαιώματα χορηγούνται μόνο στους πολίτες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτούς που έχουν την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, έτσι όπως καταλήξαμε και στη γραπτή μας απάντηση στον αναφέροντα, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν παραχωρεί εκλογικά δικαιώματα σε πρόσωπα που δεν έχουν την υπηκότητα την κοινοτική. Άρα δεν μπορεί από νομικής πλευράς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα να παρέμβει για την χορήγηση εκλογικών δικαιωμάτων στην Εστονία σε πρόσωπα που δεν έχουν την θαγένεια της Ένωσης. Αυτή είναι η απάντησή μας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριος Κάσμαν. Όχι. Η κυρία Στάνογκα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά από την Εστονία, πρέπει να πω, δεν είναι αναφορά ενός ατόμου. Συνοδεύεται από 3.000 υπογραφές. που μπορέσαμε να συλλέξουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και υπάρχει πρόβλημα ίσως με περίπου 100.000 άτομα. Δεν είναι άλλο δαπή. Πρόκειται για άτομα τα οποία διαμένουν στην Εστονία και εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα αυτής της κατάστασης. Όταν αλλοδαποί διαμένουν σε ένα άλλο κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκλογικά δικαιώματα. Δεν είναι ότι δεν έχουν το εκλογικό δικαίωμα, αλλά αυτά τα συγκεκριμένα άτομα δεν χαίρουν αυτού του δικαιώματος. Πρώτα απ' όλα στην περίπτωση της Εστονίας, για να μπορεί κανείς αυτά τα άτομα δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε εκλογές ούτε εθνικές, ούτε κοινοτικές, ούτε περιφερειακές. Και όταν μιλούμε για ευρωπαϊκές εκλογές, μιλούμε για άτομα τα οποία πρόσφατα ήρθαν στην Εστονία, αλλά μπορούν βάσει το κοινοτικού δικαίου να πάρουν μέρος στις ευρωπαϊκές εκλογές. Το θέμα είχε επανέλθει και στην Επιτροπή μας στο παρελθόν. Υπήρχαν και τέτοιου είδους αναφορές από τη Λετωνία και τώρα από την Εστονία. Και η κατάστασή τους αντικατοπτρίζεται σε δύο ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία διένυμα εγώ, συναδέλφους. Το ένα ψήφισμα είναι πρόσφατο του 2009 και αφορά την ε, ηθαγένεια την κοινοτική και λέει θεωρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ότι οι απάτριδες που μένουν μονίμως σε μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μία ιδιάζουσα θέση και α, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η πάτριδες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις περιφερειακές εκλογές. Υπήρχε και μια σχετική τροπολογία για τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά απερίφθη. Επίσης υπάρχει ψήφισμα του 2009 της δικής μας Επιτροπής που αναφέρεται στα προβλήματα που έχουν αυτά τα άτομα. Φαίνεται τώρα στις δηλώσεις της Επιτροπής ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την, ε, τους υπηκόους της Κοινωνικής Ένωσης και κάθε χώρα έχει γι' αυτό το θέμα κυρίαρχα δικαιώματα. Εμείς εφόσον κάναμε αποδεκτή, παραδεκτή αυτή την αναφορά πιστεύουμε ότι πρόκειται για παραβίαση ανθρώπινου βασικού δικαιώματος. Άρα, αν έτσι έχουν τα πράγματα, είναι θέμα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ προσωπικά επιμένω για αυτή την περίπτωση. Και χαίρομαι που ακόμη εκρεμεί αυτή η αναφορά για το θέμα αυτό. Διότι το πρόβλημα πρέπει να επιληθεί και ελπίζω ότι η Επίτροπος θα μπορέσει να μου δώσει μια απάντηση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσουμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω τη Λιθουανίας, τη Λετωνία και τη Εστονίας. Και μιλούμε για την μειονότητα που ομιλεί τη ρωσική, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως είπε η κυρία Στενόκα, η έκθεση για την παρακολούθηση μετά την ένταξη αναφέρεται στο θέμα αυτό και αναφέρεται και στους κατοίκους και το κατά πόσο μπορούν να συμμετέχουν στις τοπικές εκλογές. Υπάρχει εδώ μια ανομαλία παράξενη, ότι μπορώ να πάω στην Πολωνία και να ψηφίσω στις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά αυτοί που ζουν και πληρώνουν ε, τους φόρους τους ε, και είναι νομοταγείς πολίτες σε ορισμένε χώρες δεν μπορούν γιατί είναι απάτριδες. Το ότι έχουμε περίπου μισό εκατομμύριο απάτριδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαράδεκτο. Απολύτως απαράδεκτο. Δεδομένου ότι έχει ήδη λάβει τη θέση το Κοινοβούλιο ότι το θεωρούμε αυτό απαράδεκτο και πρέπει να επιληθεί, θα ήθελα να ζητήσω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να ζητήσουμε από τον αρμόδιο επίτροπο να στείλει μια επιστολή στην ε, κυβέρνηση να τους ζητήσει να αντιμετωπίσουν το θέμα, ιδίως ε, γιατί ε, λόγω του ψηφίσματος της 11ης Μαρτίου 2004 για την έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής για την ετοιμότητα της, σχετικά με την ένταξη διαφόρων χωρών μεταξύ άλλων και της Σλοβενίας. Συνάδελφος Στεράν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ε, είπε και η Επίτροπος ε, και ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες, ε, θέλω να πω, καταρχήν να αναφέρω το γλωσσικό πρόβλημα και μετά έχω και κάποιες παρατηρήσεις. Η αναφορά την οποία εξετάζουμε τώρα στα αγγλικά μιλάει για EP elections, στα εστονικά μιλάει για τοπικές δημοτικές εκλογές. Και θα ήθελα να ρωτήσω και τους άλλους συναδέλφους που μιλούν γερμανικά, ρουμανικά, ισπανικά. Υπάρχει αυτό το σφάλμα και στη δική τους γλωσσική εκδοχή. Στο ιταλικό κείμενο, παραδείγματο χάρη, μήπως το λάθος είναι μόνο στη δική μου γλωσσική εκδοχή. Θα ήταν απλώς μεταφραστικό σφάλμα. Αν είναι όμως σε περισσότερες γλώσσες αυτό, αυτή η διαφορετική μετάφραση, στην επόμενη συνεδρία θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Η καλή μας συνάδελφος Τατιάνα Στανόκα περιγράφει σωστά αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα των απάτριδων στην Ευρώπη είναι όντως πρόβλημα και όπως είπε ο κύριος Κάσπαν μιλάμε για μισό εκατομμύριο άτομα. Όπως είπε η Τατιάνα, η Τατιάνα είπε 100.000 αλλά είναι λίγο παλιά αυτά τα στοιχεία. Εγώ που ζω στην Εστονία το ξέρω το πρόβλημα. Δεν δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από τη Σοβιετική Ένωση το πρόβλημα. Χωρί να μπω σε λεπτομέρειε για την ιστορία, θέλω να σα πω ότι το 2003, πριν από την ένταξη στην Εστονία, είχαμε 12% πληθυσμό αυτού του τύπου. Τώρα έχουμε κατά το ίμιση λιγότερο. Μέσα σε πέντε χρόνια μειώθηκε κατά 50% αυτός ο αριθμός σε συνεργασία με τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους. Και πριν από το έτος των πολιτών το 2013 δεν θα πρέπει πια να υπάρχει καθόλου αυτό το πρόβλημα. Αύριο θα υπάρχει και μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για αυτό το θέμα. Η Εστονία έχει επιτύχει πολύ σημαντική πρόοδο επ' αυτού. Θα έλεγα εξαιρετική πρόοδο στην ένταξη αυτών των ατόμων και στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να μπορούν να ζητήσουν εστονική υπηκότητα ή αν το επιθυμούν να ζητήσουν υπηκότητα άλλων χωρών. Πράγμα το οποίο έχουν κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις και έχουμε και κάποιους Ρώσους πολίτες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους οποίους το κοινοτικό δίκαιο αρνείται το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρότι ορισμένοι συνάδελφοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι σημαντικό το θέμα και πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, εγώ θα έλεγα να το κλείσουμε το θέμα, διότι σταδιακά επιλύεται το πρόβλημα στην Εστονία. Δεν είμαι ειδικό εγώ για τη Λετωνία. Αν ε, η Τατιάνα θέλει να βάλει ένα ερωτηματικό, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι σωστό γιατί στη χώρα μου οι απάτητες μετά από πέντε χρόνια κατοικίας, μπορούν, κατοικίας στη χώρα αυτή, διαμονή στη χώρα αυτή, μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Η ετήσια μελέτη του Freedom House αναφέρει την Εστονία ως θετικό παράδειγμα σε αυτή την ε, υπόθεση και όπως σας είπα τα Ηνωμένα Έθνη θα δημοσιεύσουν αύριο μια έκθεση σχετικά με την χορήγηση υπηκότητας στην Εστονία και ε, θεωρείται επιτυχημένη η πολιτική της Εστονίας και σύμφωνα με το δίκτυ Bettelmans ε, θεωρείται τέταρτη στον κόσμο η Εστονία ως προς την πρόοδο που επιτυχάνει σε αυτά τα θέματα. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα. Και για μένα είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό. Θα το επιλύσουμε με ένα απόλυτα ευρωπαϊκό κοινοτικό τρόπο και δεν θα χρειαστεί να επανέλθουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ την Τατιάνα που υποστηρίζει τέτοιες αναφορές, γιατί τέτοιες αναφορές είναι ευπρόσδεκτες. Όπως και οι λύσεις τις οποίες περιγράφω εδώ είναι ευπρόσδεκτες. Αν ήταν πρόβλημα, και εδώ περνάω στη Λετωνία που είναι μια χώρα που δεν την ξέρω. Αν ήταν πραγματικά πρόβλημα, νομίζω ότι στη Λετωνία το κόμμα που εκπροσωπεί αυτά τα θέματα που αναφέρονται σε αυτή την αναφορά θα, είχαν και θα είχε και καλύτερα αποτελέσματα στις εκλογές. Αλλά δεν είχαν, γιατί σιγά σιγά μειώνεται η σημασία αυτού του προβλήματος όπως και στην Εσθονία, όπως σας είπα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Γιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν έχω μια ίσως αφελή ερώτηση. Ποιο είναι ο βασικό λόγο για τον οποίο δεν δίδεται η υπηκότητα, Δεν τη θέλουν, υπάρχουν κάποια άλλοι φραγμοί, κάποια άλλη αιτιολογία. Αυτοί οι οποίοι ζητούν την υπηκότητα φαντάζομαι ότι την επιθυμούν. Και λέμε ότι υπάρχουν κάποιε προποθέσει και μπορεί η απάντηση να είναι ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν ε, την ε, επικότητα. Ποια είναι η βασική αιτιολόγηση, θα ήθελα να ξέρω. Προς την ε, Επιτροπή τίθεται το ερώτημα. Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε και μαζί. Μέιερ. Ο Βίλι Μέγερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Φοβούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να στη Σοβιετική Ένωση δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να απευθυνθούμε στη Σοβιετική Ένωση για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Κατά συνέπεια, συμφωνώ με την κυρία Στάνοκα. Δηλαδή, το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό αυτή η αναφορά, διότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τέτοιου είδου προβλήματα για άτομα τα οποία γεννήθηκαν ίσως και ζουν σε μια χώρα και η χώρα αυτή τους θεωρεί απάτριδες. Μου φαίνεται λοιπόν ότι θα πρέπει όπως λέγει και η κυρία Στάνοκα, το θέμα αυτό το τρενάρουμε και από την προηγούμενη θητεία. Θα πρέπει όμως να ασκήσουμε πιέσεις ώστε να ευρεθεί μια λύση και όλοι θα πρέπει να ασκήσουμε πιώσεις. Και εμείς ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν, ώστε να βρεθεί μια λύση για αυτά τα άτομα. Ευχαριστώ, κυρίως Χάφιλτ. Νομίζω ότι η αναφορά φύγει ένα πρόβλημα που υφίσταται. Αλλά έτσι όπως είναι διατυπωμένη, δεν δείχνει και πώς θα υπάρξει λύση. Δεν πρόκειται ουσιαστικά για δικαίωμα του εκλέγην. Αλλά το δικαίωμα του εκλέγην αντικατοπτρίζει το δίκαιο περί κάθε χώρας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι ο πυρήνα. και συμφωνώ με τον Πέτερ Γιάρ και εγώ και ρωτώ, είναι σοβαρό, εδώ στο δικαίωμα ε, υπάρχουν διακρίσεις προφανείς ίσως ή κάποιοι δεν γίνονται δεκτοί ως πολίτες μιας χώρας παρόλο που εδώ και παραπάνω από μια γενιά μπορεί να μένουν νομότυπα στη χώρα. Αυτό πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που απαιτούνται και σε ό,τι αφορά τη διάρκεια χρόνου και άλλες προϋποθέσεις για να δούμε καλύτερα το θέμα. Αλλά το, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα εκλέγην, συμφωνώ και με την άποψη του εκπροσώπου της Κομισιόν ότι είναι εσωτερικό δίκαιο, οπότε το βασικό, το κέριο ζήτημα εδώ αφορά το δίκαιο περιθαγένειας. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Εστονία έχει υπογράψει τη σύμβαση σχετικά με αυτά, γιατί εμείς κάναμε μια μακρά συζήτηση όταν ε, η κυβέρνηση ξέχασε τη σύμβαση. Το θέμα αφορούσε τους ε, ανιθαγενείς Παλαιστινίους που πρέπει μεταξύ 16 και 18 ετών, τα φτάσουν σε αυτήν την ηλικία δηλαδή, να πάρουν την ε, ηθαγένεια. Είχαμε αρκετούς. Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση στη Δανία για αυτό το θέμα και η κυβέρνηση της Δανίας ε, βρέθηκε σε αμηχανία και προσπάθηκε να τα τα πράγματα και να, βέβαια, να τα αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Είναι σημαντικό να ξέρουμε αν έχει η Εστονία υπογράψει τη σύμβαση, γιατί αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι γεννήθηκαν στην Εστονία, Όταν φτάσουν στην ηλικία των 18 ετών, αυτομάτως, αν ζητήσουν την ηθαγένεια, ε, ε, τους χορηγείται. Αυτό είναι μία πλευρά του ζητήματος. Αν έχετε υπογράψει τη σύμβαση, έτσι πρέπει να γίνεται. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει πάντα προσπάθεια να μειώνεται ο αριθμός των ανηθαγενών. Αυτός είναι ένας βασικός σκοπός. Οπότε να βρεθεί μια ηθαγένεια για όλους αυτούς τους ανθρώπους. δεν θυμάμαι πώς τη λένε τη σύμβαση αυτή, αλλά είναι πολύ ε, σημαντική. Υπάρχει και συζητήθηκε στη Δανία έντονα. Δεν γνωρίζω την δίκη, αλλά άκουσα τι είπατε. Αν κάποιος όμως έχει γεννηθεί πριν από 5 χρόνια, θα γίνει 18. Ούτως, ούτως ή άλλως τα 18 παίρνει την υπηκονότητα. Εμείς είμαστε λίγο μπροστά, μπροστά από τις... Δεν ξέρω ότι χρειάζεται να ζητήσουμε άλλη απάντηση από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για αυτή την αναφορά. Δεδομένου ότι όπως είπαμε χάρη στην κυρία Ζάνοκα θα το θέμα στην Επίτροπο και πιστεύω ότι θα περιμένουμε τη γραπτή απάντησή της βάσει της οποίας θα κάνουμε ενδεχομένω περαιτέρω συζήτηση. Πιστεύω λοιπόν ότι παραμένει η αναφορά αυτή ανοιχτή και θα περιμένουμε την απάντηση δεδομένου ότι ασχολείται προσωπικά με το θέμα αυτό η κυρία Ρέντινγκ. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Μια ερώτηση σύντομα που ενδιαφέρει την Επιτροπή, όχι σε σχέση με την Κομισιόν. Αν αληθεύει αυτό που είπε πριν από λίγο ο συνάδελφος Τέρενς, ότι δηλαδή υπάρχουν προδιαγραφές, προϋποθέσεις που σε ένα αποφασιστικό νομικό ερώτημα ε, παρουσιάζουν αποκλήσεις, εδώ υπάρχει θέμα. Βέβαια δεν μπορούμε εμείς τώρα να το τσεκάρουμε αυτό το θέμα. Παρακαλώ λοιπόν κατά εξαίρεση να ελέγξει τις μεταφράσεις η γραμματεία και αν υπάρχουν διαφορές να μας εξηγήσει γιατί. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Τι πρόκειται, τι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή τις δημοτικές. Αυτό είναι κεντρικό ζήτημα για όσους ξέρουν τα συνταγματικά ζητήματα, οπότε πρέπει να διευκρινιστεί. Σίγουρα θα τα ελέγξουμε και θα δούμε τις ε, μεταφράσεις στις διάφορες γλώσσες και αν ευθυγραμμίζονται ε, σε αυτή την αναφορά. Λοιπόν, το τελευταίο, ο κύριος Μάιερ ε, είναι ο εισήγητης για την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής των Αναφορών. Θέλετε λοιπόν να αρχίσετε τη συζήτηση, να κάνετε μια εισαγωγή. Φύγε, φύγε. Σήμερα το πρωί μου Είναι πολύ γρήγορα τα πράγματα λοιπόν. Ούτω ή άλλω θα ήθελα να καλέσω του συναδέλφου όπω κάθε χρόνο η ετήσια έκθεση να είναι το αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας και να προσπαθήσουμε στην έκθεση αυτή να συμπεριλάβουμε όλες τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων για να μπορέσουμε να κάνουμε απολογισμό της εργασίας μας κατά τη διάρκεια του 2010 στην Επιτροπή Αναφορών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιέχει μια ένα συγκεκριμένο περιγραφικό μέρος για να πούμε τι ακριβώς κάναμε το 2010. Να αναφέρουμε τον αριθμό των αναφορών, ανακράτω το ποσοστό των θεμάτων που επιλύσαμε, αυτές που παραμένουν ανοιχτές, τέλος πάντων μια πολύ περιγραφική ετήσια έκθεση και να είμαστε σε θέση με γενικό τρόπο να δούμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία χειριστήκαμε από αυτά τα οποία που απασχολούν τους πολίτες μας, να παραθέσουμε κάποια παραδείγματα ξένων των πολιτικών ομάδων και τελικά να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια διδακτική έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι ελλείψεις, οι αδυναμίες που έχουμε τη στιγμή που καλούμεθα να δώσουμε μία αποτελεσματική και γρήγορη απάντηση στους πολίτες και από την άλλη να σημειώσουμε πόσο καλή δουλειά έγινε και πού καλή, έγινε καλή δουλειά στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να καλέσω τους και τις συναδέλφους το συντομότερο δυνατό να ορίσουν αυτός ο οποίος θα ε, παρακολουθήσει αυτή τη δουλειά για να μπορέσω εγώ να ολοκληρώσω την εκθεσή μου και να την παρουσιάσω έγκαιρα. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κανείς το λόγο? Όχι, δεν βλέπω κανένα να θέλει το λόγο. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε όλα τα θέματα της μερικής διάταξης. Για το τμήμα Β δεν έχει κάνει κανείς ε, κανένα σχόλιο. Μάλλον λάθος. Έχουν γίνει δύο παρατηρήσεις από τον κύριο Μάγερ για το τμήμα Β. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τα δύο αιτήματα. Λοιπόν, εγκρίνεται ο κατάλογος με τις τροπολογίες που πρότεινε ο κύριος Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ.